Λοιπόν, εντάξει, Τρίτη, ναι. έξι, το απόγευμα. Ευχαριστώ τον κύριο Τρισέ για τη συμμετοχή του σε αυτόν τον νομισματικό διάλογο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε επί ιονή θεσμικής βάσης. Θα σας υπενθυμίσω τα δύο θέματα, τα οποία είχαμε προτείνει για αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τρισέ. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν θέλετε, του αποπληθωρισμού ή του στάσιμου πληθωρισμού, και πώς θα μπορούσαμε να αναδιαρθρώσουμε την ε, διεθνή χρηματοοικονομική δομή. Παρακαλώ κύριε Τρισέ να μιλήσετε για 10 λεπτά και κατόπιν θα ακολουθήσει αυτό το οποίο γνωρίζετε απ' έξω και ανακατοντά. Ο κύριος Τρισέ λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη Κυρίε και κύριοι μέλη τη Επιτροπής, με μεγάλη μου χαρά έχουμε αυτή την ε, πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή του 2009 ε, λίγες μέρες μόλις μετά από την συνεδρίαση του Διοικητικού μα Συμβουλίου στις 15 Ιανουαρίου για την νομισματική πολιτική επίσης την Τρίτη στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα κατά την ε, Ολομέλεια στην πανηγυρική συνεδρίαση για τα 10 χρόνια του ευρώ μεγάλη μου χαρά ε, διαπίστωσα ότι είσαστε αναφανδόν υπέρ του ευρώ και της κεντρικής τράπεζας. Ξεκινώ με μια αξιολόγηση της οικονομικής και νομιματικής ε, συγκυρίας και θα σας εξηγήσω τους λόγους στους οποίους βασίστηκαν οι αυτές οι πρόσθετες αποφάσεις μας για τα επιτόκια. Θα ήθελα να πω ε, κάτι το οποίο αναφέρεται στα, στην Ευρωζώνη και στο τέλος θα ήθελα να απαντήσω σε θέματα της, ε, του ε, διεθνούς χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος. Το θέμα αυτό κατά τους επόμενους μήνες αναμφίβολα θα αποκτήσει και μεγαλύτερη σημασία. Uh, Πρώτα για τι οικονομικέ νομικέ εξελίξει, από τότε που τα είπαμε για τελευταία φορά στι 8 ε, Δεκεμβρίου, η οικονομική συγκυρία, το οικονομικό κλίμα συνεχίζει να επιδεινώνεται και έχουμε επίση και συρρήγνωση του ρυθμού του πληθωρισμού. Το Δεκέμβριο του 2008 το, ο πληθωρισμός έτρεχε με 1,6% και επίση οι πληθωριστικές πιέσει και οι κίνδυνοι έχουν από τότε μειωθεί και αν κοιτάξουμε στο μέλλον όπως πρέπει με μια προοπτική μεσοπρόθεσμη για την οικονομική πολιτική και να λάβουμε υπόψη και τις αποφάσεις μας και και την τελευταία απόφαση για την οικονομική πολιτική θα δούμε όσον αφορά την Ευρωζώνη ότι ο πληθωρισμός ευθυγραμμίζεται με την πολιτική μας για την σταθερότητα των τιμών όσον αφορά τον ορίζοντα της οικονομίας πολιτισμικής και μεσοπρόθεσμα ε, ε, έτσι ε, αποφάσισαν οι οι διοικητέ των τραπεζών. Από το Σεπτέμβριο είχαμε αυτή την κρίση, έχουμε εντάσεις οι οποίε χτύπησαν και την πραγματική οικονομία και επίση θα πρέπει να ρίξουμε ματιά τι γίνεται με την ζήτηση σε παγκοσμίο επίπεδο, τι γίνεται στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε ότι τα πράγματα θα είναι κατάσταση ύφεση για μια μεγάλη περίοδο. Επίση, ο μειωμένο πληθωρισμός ε, θα βοηθήσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και άρα η, στην Ευρωζώνη η οικονομία θα ωφεληθεί από αυτά τα πάρα πολύ γενναία και μακρόπονα μέτρα οικονομικής πολιτικής που τις τελευταίες εβδομάδες αποφασίσαμε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κλίμα αυτό χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα, υπάρχουν κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη και επίσης αυτό έχει να κάνει και με τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην πραγματική οικονομία. Αλλά επίσης υπάρχουν και ανησυχίες σε σχέση με το ε, ότι μπορεί ξαφνικά να εμφανιστούν και να ενταθούν ε, μέτρα και πιέσεις ε, προστατευτισμού. Γιατί μπορεί να έχουμε υπερδιόρθωση του ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποια βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να λάβουν τι ευθύνε του. Άρα, θα πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και να έχουμε μια προοπτική μεσοπρόθεσμη στη μακροοικονομική μας πολιτική και έτσι να έχουμε μια προσέγγιση ε, προσδοσμένη προς σταθερότητα και αυτό είναι το καλύτερο για να μπορέσουμε να ε, δώσουμε αξιοπιστία στην οικονομία χρειάζονται επομένω κάποια μέτρα από τις κυβερνήσεις εναντίον της κρίσης για να ξαναυπάρξει εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και έτσι να χαλαρώσουν οι, οι πιέσεις όσον αφορά τις πιστώσεις προς ε, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τελευταία στοιχεία μας δείχνουν ότι έχουμε <clears throat> αναζωπήρωση ε, ε, στο νομισματικό, στην νομισματική πολιτική και η Δέκεντρική Τράπεζα είπε ότι θέλει ο πληθωρισμός να είναι πολύ κοντά στο 2% λίγο πιο κάτω. Έτσι θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες για σταθερότητα. Και την περασμένη εβδομάδα αποφασίσαμε να μειώσουμε το επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης και να πάμε στο 2%. Και έτσι η συνολική μείωση από τον Οκτώβριο του 2008 έφτασε στα 225 ε, μονάδες βάσης. Και τώρα, για να δούμε περισσότερο τον ορίζοντον μέσο πρόθεσμο όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών στην Ευρωζώνη. Κυρίως να δούμε τι γίνεται με τη διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού όπως τώρα ε, παρατηρούμε να συμβαίνει. Και θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ συγκράτηση του πληθωρισμού και αποπληθωρισμού. Συγκράτηση του πληθωρισμού σημαίνει να συγκρατείται ο ρυθμό του πληθωρισμού. Κάτι το οποίο προέρχεται από οικονόμηση δαπανών όσον αφορά την προσφορά λόγω αποτελεσματικότερης άσκηση του εμπορίου. Κάτι το οποίο πολλέ φορέ συνοδεύεται από ξαφνικά χτυπήματα αρνητικής ζήτησης όπως γίνεται τώρα. Όμως ε, είναι κάτι θετικό αυτό το φαινόμενο και αυτό διότι έτσι υποστηρίζεται, βοηθάται το πραγματικό εισόδημα στη σημερινή συγκυρία βλέπουμε να υπάρχει μετεσυγκράτηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Κυρίω αυτό προκύπτει από μια απότομη μείωση των τιμών καυσίμων και εμπορευμάτων. Οπότε γι' αυτό και λέμε ότι είναι θετική εξέλιξη. Η απότομη άνοδος που είχαμε για στο πετρέλαιο και στα εμπορεύματα ξεκίνησε το 2007 και έφτασε μέχρι τα μέσα του 2008. Ε, αυτό είχε πληθωριστικό χαρακτήρα και χαρακτήρα τη οικονομίας. Όμως έτσι με το που τόσο πέσαν αυτές οι τιμές αυτό μας οδηγεί σε τέτοιου είδους ε, φαινόμενο συγκέντρωση του πληθωρισμού αλλά και αυτό είναι και μπορεί να οδηγήσει σε κάτι θετικό για την οικονομία 15,4% ε, είχαμε τη μείωση της τιμής του καυσίμου και αυτό σημαίνει στο καλάθι για τον πληθωρισμό 5% στο δίκτυο τιμών μάλλον Βλέπουμε επομένω ότι οι εξελίξει όσον αφορά την προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντικέ και βλέπουμε ότι επίση η συγκέντρωση του πληθωρισμού μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αρνητικά νούμερα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τι προσδοκίε μα ε, για τον πληθωρισμό σε έναν ορίζοντα μέσο πρόθεσμο. Όμω από την άλλη μεριά, ο Αποπληθωρισμό είναι μία διαρκή και αυτοτροφοδοτούμενη μείωση ε, μιας μεγάλης βεντάλιας τιμών αυτό είναι ένα κυκλικό φαινόμενο το οποίο το, φέρνει, το φέρνουν κάποιες τιμές οι οποίες πέφτουν και υπάρχει προσδοκία να πέσουν περισσότερο. Έτσι η συγκράτηση της ζήτησης συνεχίζεται οπότε ε, ε, έτσι, έτσι συνεχίζεται η πίωση στις τιμές για περαιτέρω πτώση. Δεν κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο τώρα. αυτή τη στιγμή ακριβώς οι προσδοκίες ε, πληθωρισμού που έχουμε είναι η καλύτερη άμυνά μας τόσο ώστε να μην φτάσουμε σε τέτοια κυκλικά φαινόμενα ε, πληθωρισμού. Και γι' αυτό σας λέω ότι έτσι βλέπετε ότι τώρα έχουμε μια κατάσταση συγκράτησης του πληθωρισμού το οποίο ε, έχει τις ρίζες του σε αυτήν την πάρα πολύ σημαντική μείωση τιμών ψήμων και εμπορευμάτων. President, namely the international financial architecture. I consider that the fragility... Για να δούμε τώρα πώς έχει η χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική παγκοσμίω. Βλέπουμε ότι υπάρχει, το, το, το, σύστημα έχει γίνει πάρα πολύ ευάλωτο. Είδαμε τώρα η κρίση πώς χτύπησε το σύστημα, κάτι που είναι απαράδεκτο. Άρα θα πρέπει να αντλήσουμε ό,τι συμπέρασμα ήταν από την κρίση, ε, να σταματήσει κάθε αυταρέσκεια και να λάβουμε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία του στήματος θα πρέπει να βελτιωθούν. Τη διαχείριση του κινδύνου, η διαχείριση της ρευστότητας, ε, η άμυνα ε, των, του, του ιδιωτικού, ναι, των ιδιωτικών ιδρυμάτων, η διαφάνεια των αγορών και το κατανοητό των χρηματοπιστωτικών μέσων. κάνατε και εσείς κάποιες δημόσιες ακροάσεις και καταλήξατε κι εσείς ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Ε, θα πρέπει να αφήσουμε τα συμφέροντα ε, στην άκρη και επίσης να μην βλέπουμε το βραχυπρόθεσμο κέρδος και επίσης θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους αποτελεσματική άμυνα στα κυκλικά φαινόμενα ε, που πολλές φορές δημιουργούνται από το όλο το πλέγμα των κανόνων που έχουμε για τα λογιστικά και γενικά για το κανονιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να έχουμε τον δυναμισμό ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τα συμφέροντα όπου υπάρχουν και το G20 αλλά και το Διεθνές Ταμείο είναι αποφασισμένοι να δράσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως για να λειτουργήσουμε ε, αποτελεσματικά δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται επίσης κάποια στιβαρή πολιτική μακροοικονομική ε, με ορίζοντα μέσο και μακροπρόθεσμο να αποφύγουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έλλειψη ισορροπιών κάτι το οποίο θύνεται κατά πολύ για την σημερινή κρίση. Επίσης χρειάζεται υποπτή αποτελεσματική των μακροοικονομικών πολιτικών για τις, και αυτό αφορά τις ε, συστημικές πλευρές του, των οικονομιών. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το νομισματικό Ταμείο και γι' αυτό και θα πρέπει η εντολή του να ενισχυθεί. Απλώ θεσμική τώρα. Μπορούμε να έχουμε τις εξή βελτιώσεις. Πρώτα-πρώτα, η αρχιτεκτονική του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, χρηματοπιστωτικού συστήματος, χρειάζεται να ενισχυθεί μέσω του Financial Stability Forum και του G20. Το Financial Stability Forum είναι μοναδικό, γιατί εκεί είναι ένα βήμα για όλα τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τις αρχές που συστημικά δρούν επί των αγορών. Δεν έχει και τον καθημερινό χαρακτήρα και είναι και ανεξάρτητα από πλευράς πολιτικής. Πρέπει να διευρυνθεί όμως αυτό το, το, όργανο, αυτός ο θεσμός και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που έχουμε αυτή την ε, συγκυρία και αυτό αφορά και το G20 χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και το G7 ε, δεν ε, χρησιμεύει άπαξ και η σημερινή κρίση πήγασε από τις βιομηχανικά προηγμένες κοινωνίες και χώρες δεύτερον όσον αφορά την εντολή του νομισματικού ταμείου θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι πιο αποτελεσματική η διοίκησή του, το ίδιο αφορά και την Παγκόσμια Τράπεζα, πώς θα είναι πιο πλήρης εκπροσώπηση εκεί των αναδειωμένων ε, οικονομιών αντίστοιχα με την σημασία τους για την παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι κάτι το απαραίτητο. Ε, κατακλείδη, να σας τονίσω δύο τεινά. Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα, όσον αφορά τις πολιτικές στην Ευρωζώνη, Υπάρχουν εδώ πέρα διαφοροποιημένοι ρυθμοί ε, αύξησης των μισθών. Έτσι έχουμε αποτελεσματικότητα διαρθρωτική. Δεν έχουμε ευθυγράμμιση εθνικών πολιτικών. Αυτό μας κοστίζει σε ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων και άρα θα πρέπει να κάνουν διαρθρωτικές, μετα... μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν αυτό που χάθηκε σε ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται συγκράτηση των τιμών, αλλά και των μισθών. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο θέλει να τονώσει τα δημοσιονομικά με αντίστοιχες φορολογικές πολιτικές. Να χρησιμοποιηθεί κάθε περιθωρισμό που προσφέρει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει η αύξηση του δημοσίου χρέους όμως ταυτόχρονα και με τις ενέργειες στο φορολογικό να οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης εκ μέρους του κόσμου στην οικονομία. Γιατί έτσι θα εκμηδενήσουμε τις ωφέλειες από αυτή τη νέα πολιτική. Για να δούμε τώρα ε, τι μπορούμε να πούμε για την ε, εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Χρειάζεται κάτι να ρυθμιστεί σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την Ευρώπη τώρα χρειάζονται κάποιες μακρόπνες λύσεις. η ομάδα υψηλού επίπεδου του Ζακ Ντελαροζιέρ πρόκειται να υποβάλει κάποιε προτάσει και αυτό φαντάζομαι θα συμβάλλει πάρα πολύ στο να δημορφώσει πολιτική μα. Και εσεί άλλωστε θα τα συζητήσετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να λύσει έχουμε. Έχουμε το άρθρο 105 παραγράφος 6 συνθήκη το οποίο ορίζει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Κινητική Τράπεζα συγκεκριμένες ε, ενέργειες όσον αφορά την εποπτεία του γνωτοπιστωτικού τομέα. Ήδη έχει αρχίσει η διαβούλευση όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει η Κεντρική Τράπεζα και το δικό της Συμβούλιο. Σε αυτή την φάση πάντως ακόμα δεν έχει προκύψει κάποια απόφαση. Όταν έχουμε κάτι θα σας αναφέρουμε σχετικώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τρισέ. Το άρθρο 105, σημείο 6 τη συνθήκη, δίδει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωμα έκφρασης και γνώμης. Θα είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί παρατηρητές. Σύμφωνα με τους κανόνες θα δώσω το λόγο στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Και καταρχήν στο ΕΛΚΑ. Για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία σημεία. Να σας απευθύνω τρεις ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στι τελετέ για την δεκάτη επέτειο του ευρώ στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Και οι τίτλοι στον τύπο είναι θα εκραγεί το ευρώ με την κρίση. Θα πρέπει συνεπώς να περάσει ένα ισχυρό μήνυμα που θα αποφύγει τέτοιου είδου στήρες και άκαρπες συζητήσεις. Δεύτερον, Διάβασα με μεγάλο ε, ενδιαφέρον ε, στην παρέμβασή σας στο Συμπόσιο των Παρισίων στις 19 Ιανουαρίου για τους κινδύνους στη χρηματοοικονομική αγορά. Θα μπορούσατε να μας πείτε, αν κατά τη γνώμη σας, πού είναι ε, το αίτιο, πού βρίσκεται η αιτία αυτής της τύφλωσης, ας το έτσι. Και τελευταία ερώτηση. Σήμερα έχουμε υπάρξει εγκλωρισμό όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων παρά τι προσπάθειε που κατέβαλε η ΕΚΤ και τα κράτη-μέλη. Δεν διανέμονται τα κονδύλια. Και αυτή αποτελεί μια σοβαρή δυσκολία για την οικονομία, για τι επιχειρήσει και ειδικότερα για τι ΜΜΕ. Ποιε είναι κατά τη γνώμη σα οι δυνατότητε να έχουν άμεση εφαρμογή τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν και θα φέρουν αποτελέσματα επίση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρωβουλευτά για τις τρεις αυτές σας ερωτήσεις. Για το πρώτο σας ερώτημα. Θα σας έλεγα ότι εννοείται και εξυπακούεται ότι η ευρώ και η ευρωζώνη έδειξαν αντίθετα την ε, ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτή την κρίση. Την οποία παρατήρησαν αυτό και όλοι οι παρατηρητές. Και όλα τα νομίσματα του κόσμου βρίσκονται υπό την πίεση της παρούσης συγκυρίας και των οικονομικών αυτών διαταράξεων και θα έλεγα όλα τα νομίματα του κόσμου χωρίς καμία εξαίρεση πρέπει να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία. Το ίδιο ισχύει για όλα τα νομίσματα με τα οποία έχουμε σχέσεις εμείς. Αυτό ισχύει για τη στελίνα, το δολάριο και για όλα τα λοιπά νομίσματα. Θα έλεγα λοιπόν ειλικρινέστατα ότι οι παρατηρήσεις αυτές τις οποίες διατυπώσατε μου φαίνονται εντελώς αβάσιμες και βεβαίω θα πρέπει να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε ε, το μέτρο του δυνατού από δική μα πλευρά στην νομισματική πολιτική, το ευρώ δηλαδή, και το, οι κυβερνήσει δηλαδή να εφαρμόσουν τη δική του νομισματική πολιτική, διότι είναι υπεύθυνε αυτέ τι κυβερνήσει για τη ε, πολιτική διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων, για την συγκράτηση του κόστου, όπω επίση και την δημοσιονομική πολιτική. Για το δεύτερο σα ερώτημα τώρα. Νομίζω ότι Περάσαμε και άλλα επεισόδια πριν να ξεκινήσουν αυτές οι οικονομικές διαταράξεις τον Αύγουστο του 2007. Υποτίμησης τόσο του όγκου των κινδύνων στην διεθνή οικονομία και του τιμήματος και αυτό υπόθηκε δημόσια και κατά επανάληψη και πληστάκες από πολλούς μεταξύ των οποίων και των κεντρικών τραπεζών και εγώ ο ίδιος το είπα αυτό ως πρόεδρος και ως Προεδρεύων της ομάδας των 10 κεντρικών και του Global Economy Meeting στο οποίο συναντώμε με τους συναδέλφους μου και τους ομολόγους μου για να δούμε τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας είπαμε ότι υπάρχει αυτή, υποτιμήθηκε αυτή η κίνδυνη τελικά και οι λόγοι είναι πολύ άριθμοι δεν υπάρχει μόνο ένα αίτιο πολλά ότι είναι πολύ εξελιγμένα αν θέλετε, τα χρηματοοικονομικά αν θέλετε, μέσα και εργαλεία. Γι' αυτό και επιμένω στην απαραίτητη διαφάνεια. Υπήρξε η έκρηξη επίση κάποιων αγορών, οι οποίε οι ίδιε δεν παρουσίαζαν διαφάνεια και διευκόλυνα την ανάληψη του είδου περίγων κινδύνων. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι μακροοικονομικοί παράγοντε διεθνώ, η αύξηση τη τιμή του πετρελαίου δηλαδή και των πρώτων υλών που οδήγησε σε αναγκαστική αποταμίευση σε διεθνές επίπεδο και οδήγησε ένα μεγάλο αριθμό επενδυτών στην συστηματική αναζήτηση υψηλών αποδόσεων, υψηλών κερδών, άρα και υψηλών κινδύνων. Το αν λέω όλα αυτά και δεν καλύπτω τα πάντα, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι. Όπω επίση και ότι, ότι τυφλώθηκαν των εισαγωγικών, αν θέλετε, εκείνοι που συμμετέχουν σε αυτέ τι αγορέ δηλαδή και οι εμπλεκόμενοι φορεί. Είναι πολυδιάστατοι αυτοί οι λόγοι, πολυδιάστατοι. Γι' αυτό λοιπόν που επιμένω ότι θα πρέπει να μεταρρυθμίσουν τα πάντα. Να μην αφήσουμε τίποτα στη σκιά και εκτό. Να μην εφαρμόσουμε και να ακολουθήσουμε πολιτική, την πολιτική του αποδιοπομπαίου τράγου, γιατί αυτό θα μα αναγκάσει να εστιάσουμε τη ζωή μα σε ορισμένου μόνο παράγοντε αυτή τη κρίση και όχι σε όλου. Θα πρέπει συνεπώ να τα δούμε όλα αυτά εκ του σύνεγγυ και να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Και κατόπιν έχουμε και αυτό το μείζον ερώτημα τη συνήθου και τη φιλολογική λειτουργία τη οικονομία έγιναν και κατευλήθηκαν σημαντικέ ε, προσπάθειε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι λοιπέ κεντρικέ τράπεζε, από τι κυβερνήσει έγιναν δηλαδή. Με προθυμία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό την παρούσα συγκυρία, δεν είμαι βέβαιο. Βεβαίω ότι το σύνολο όλων των εμπλεκομένων φορέων έχει καταλάβει και έχει αντιληφθεί δηλαδή το τι έχει ακριβώ γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται, επαναλαμβάνω. Γιατί θα πρέπει ε, να είμαστε υπό επαγρύπνηση, συνεχή, διαρκή όλοι εν πάση πτώσει οι οικονομικοί παράγοντες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό ισχύει βεβαίως για τις τράπεζες, όλος ιδιαίτερος. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μίτσελ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τρίσε, φαίνεται ότι ε, το κλίμα των επιτοκίων πρόσφατα διαμορφώνεται πολύ συγκρατημένα. Όμως ε, ευτυχώς ε, έχουμε έναν θεσμό που μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Αναφέρατε στις παρεμβάσεις σας ότι το να επανέλθει η εμπιστοσύνη αυτό είναι κλειδί στην όλη υπόθεση. Οι τράπεζες μοιάζουν να έχουν εμπιστοσύνη μία στην άλλη και πώς ακριβώς εμφανίζεται αυτό στα διατραπεζικά επιτόκια. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να καταστεί ένα στοιχείο κλειδί ε, στην πολιτική σας. Μιλήσατε ε, αυτό το μήνα νομίζω για την ανάκαμψη και χαίρομαι που μιλήσατε για την ανάκαμψη. Είναι πλέον η στιγμή να, να μιλάμε για την ανάκαμψη. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτήν. Και αν δεν μιλάμε δεν θα έρθει. Ε, επίσης, ε, ε, να ε, μιλάμε για το πώς προτιθέμεθα να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτή την ε, ανάκαμψη σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Ναι, να διαχειριστούμε την κρίση, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε και ένα όραμα του τι θα συμβεί όταν θα έρθει η ανάκαμψη και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να έρθει πολύ. Όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι τράπεζες καταρχήν πρέπει να αρχίσουν να δείχνουν εμπιστοσύνη η μία στην άλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, να πω το εξής. Όπως είπα και παλαιότερα εδώ στις ακροάσεις εξετάζουμε πολύ προσεκτικά την ε, λειτουργία των ε, αγορών χρήματος και έχουμε πει επανειλημμένα ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει πολύ προσεκτικά το Euribor και κυρίως ε, το ότι υπάρχει μεταφορά των δικών μας των αποφάσεων για την νομισματική πολιτική στα επιτόκια που τελικά ε, ισχύουν στην αγορά χρήματος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι αυτό που διαπιστώσαμε τις ε, τελευταίες εβδομάδες όσον αφορά το Oribor, το τριμηνιαίο επιτόκιο, σωστή είναι η κατεύθυνση που ακολουθειτε Δηλαδή βλέπουμε σιγά σιγά ε, το επίπεδο των επιτοκίων αυτών να κατεβαίνει όλο και πιο κοντά ε, προς το δικό μας το όραμα του τι πρέπει να είναι ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι πιο κοντά στις ε, πολιτικές μας. Έτσι λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα βλέπω να υπάρχει κάποια βελτίωση στην αγορά χρήματος. Πρέπει όμως να επαγρυπνούμε Ευχαριστούμε ε, ουσιαστικά και να ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν τα πάντα όπως θα έπρεπε με την έννοια ότι για αρκετούς λόγους εξακολουθεί να υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα ανάμεσα στις ίδιες τις τράπεζες οποτεδήποτε ε, έχουν συναλλαγές. Όσον αφορά όμως το δίκτυ του Euribor που τον παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά πράγματι έχει σημειωθεί πρόοδος και ε, θέλουμε η πρόοδος αυτή να συνεχιστεί. Όσον αφορά το χρόνο που θα επέλθει η ανάκαμψη και εγώ ο ίδιος είπα ότι ε, πράγματι θα υπάρξει ανάκαμψη αλλά σας είπα και πριν ότι το επίπεδο της ανασφάλειας ε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό αφορά όλους τους θεσμούς ε, εθνικούς ή διεθνείς. Μετά το 2009 όπου θα είναι και είδαμε ένα έτος που προηγήθηκε ύφεσης Θέλουμε το 2010 να είναι ένα έτος όπου θα έχουμε και πάλι θετικές εξελίξεις, μια χρονιά που θα ακολουθήσει μετά από δύο δύσκολες χρονιές, το 8 και το 9. Αυτή η παρατήρηση νομίζω ότι μπορεί να γίνει για την οικονομία της ε, Ευρωζώνης και νομίζω ότι μπορεί και να λεχθεί γενικότερα για την ε, παγκόσμια οικονομία. Ε, συζητάμε με τους ε, προέδρους όλων των άλλων ε, σημαντικών οικονομιών και των αναδειωμένων και έχω την εντύπωση, επικρατεί η αίσθηση ότι το 2010 θα μπορούσε να είναι η χρονιά έναρξης ανάκαμψης ε, της οικονομίας γιατί τώρα πλέον έχουμε συντονιστεί όλες οι οικονομίες του κόσμου συμπεριλαμβανομένων και των αναδειωμένων Σύμφωνα με αυτά που είπατε. Πράγματι υπήρξε μία τεράστια υποτίμηση του όγκου και του κινδύνου κατά τα προηγούμενα έτη και αυτό είναι η ρίζα του κακού, το αίτιο των αναταραχών που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως αυτό θα ε, μπορούσε και να οδηγήσει και στο να υποτιμήσει κανείς τη δυνατότητα της παγκόσμιας οικονομίας να ανακάμψει. Γιατί στην περίπτωση αυτή πολλοί θεσμοί και οι δυτικοί θα μπορούσαν να χάσουν την ευκαιρία να είναι παρόντες τη στιγμή που θα αρχίσει η ανάκαμψη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι όλοι συλλαμβάνουν αποφάσεις διοικητικά συμβούλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να έχουν τεντωμένες τις κεραίες τους. Παρατηρούμε τώρα την τιμή ε, του πετρελαίου των βασικών αγαθών της ενέργειας. Οι τιμές αυτές είναι πολύ πιο χαμηλές, όπως είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Βεβαίως και είναι αυτό αποπληθωριστικό. Αλλά αν θέλετε, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση είναι ε, ανακαμπτικό ας το πούμε έτσι το στοιχείο και αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί τελικά θα υπάρξει ανάκαμψη. Ε? Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η πίστη με επικεφαλαίο στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Ο κύριο Σαλμούνια, ο επίτροπο Σαλμούνια μα είπε ότι χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή ελάχιστοι δημόσιοι κρατικοί πόροι. Πολλέ ε, τράπεζε προτιμούν να καταθέτουν, να βάλουν τι καταθέσει του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρά να την επενδύσουν στην πραγματική οικονομία τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Μιλήσατε κατόπιν ε, την, ε, για την οδηγία για τις κεφαλιακές απαιτήσεις. Και ακούστηκε από ενό κοινό ότι αυτό δεν θα βοηθούσε στην επίλυση των προβλημάτων. Γιατί θα οδηγούσε, αν θέλετε, σε κάποια προκυκλικά φαινόμενα. Τώρα η Fed κάνει δάνεια τριετούς διάρκειας. Πολλοί πιστεύουν ότι θα έπρεπε να, την, ε, να το αυξήσουμε αυτό το χρονικό όριο διότι εκείνοι οι οποίοι αν θέλετε θέλουν να δανείσουν περισσότερο μακροπρόθεσμα να έχουν και τη βεβαιότητα ότι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποιο κέρδος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς παρατηρούμε και διαπιστώνουμε και συνδέεται με το γεγονός ότι Θέλουμε πάση θυσία να αποφύγουμε κινδύνου συστημικής ρευστότητα. Γι' αυτό λοιπόν παρέχουμε ρευστότητα επί περίοριστου βάσους σε εμπορικές τράπεζες στην Ευρωζώνη μια εβδομάδα, για ένα μήνα, τρει μήνες, έξι μήνες. Επ' αυτή τη βάσεω ή επ' αυτών των βάσεων. Και αυτό συνδέεται επίσης, όπως ε, αναφέρθηκε και από τον προηγούμενο μιλητή, στο γεγονό ότι οι τράπεζε οι ίδιε τίνουν ναι, παρόλο που η χρηματική αγορά αν θέλετε αρχίζει να παρουσιάζει μια αναζωγόνηση την ρευστότητα της κεντρικής τράπεζας στην παίρνουν και όταν υπάρχει έξα ρευστότητα τότε αν θέλετε την καταθέτουν σε αυτό το deposit facility κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ζωγονίσουμε ούτως υπήν την, ε, αυτές τις αγορές παρατηρούμε τα τριμηνία Euribor που δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η προοδευτική ε, η σταδιακή αναζωγόνηση της αγοράς ή των αγορών και αποφασίσαμε πρόσφατα και αυτό το μέτρο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και να λειτουργεί να διευρύνουμε θέλει τον διάδρομο που έχουμε που είναι ένα επιπλέον εργαλείο που έχουμε στην διάθεσή μας για να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση ούτως υπήν της, ε, των χρηματαγορών. Επίσης, όσον αφορά το άλλο σας ερώτημα, πρέπει να υποθεί ότι δεν αποτελεί πρόθεση υπό την παρούσα κατάσταση. Δεν υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσει. Δηλαδή αυτό θα αποτελούσε προκυκλικό φαινόμενο. Και είπα ότι θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή την προκυκλικότητα. Εν πάση περιπτώσει και πιο συγκεκριμένα επί την παρούσα συγκυρία. Θέλουμε να φτιάξουμε αυτά τα buffers, αυτούς τους προφυλακτήρες επιπλέον ε, και πρόσθετα ως προς τις κεφαλαϊκές απαιτήσει για να μπορέσουν ε, να καλύψουν ε, τις απώλειες τις οποίες θα υποστούν στο μέλλον. Δεν μιλούμε δηλαδή για αύξηση και των κεφαλαϊκών αποτήσεων, αλλά μια συνετή προσέγγιση να έχουμε αυτούς τους προφυλακτήρες σε περίπτωση που θα χρειαστούν αλλά το ερώτημά σας ήταν πολύ εύστοχο και είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Παρουσία αυτών των εντάσεων, αλλά και στο μακροπρόθεσμο μέλλον, να αποφύγουμε αυτή την προκυκλικότητα ως προς τη ε, συμπεριφορά μας και τις αντιμετωπίσεις μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Τράπεζα, εμείς παρέχουμε ρευστότητα επί εβδομαδιαίας, μηνιαίας, τριμηνιαίας, ξεμηνιαίας βάσεως, επί απεριορίσου βάσεως, πρέπει να βελθήσουμε όσο μπορούμε την αγορά να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει καλύτερα όμως αυτή τη φορά. Και βλέπουμε κάποια στοιχεία εδώ. Αρχίζουμε ότι η σταδιακή, αν θέλετε, προοδευτική βελτίωση υπάρχει, αλλά θα πρέπει, όπως σας είπα προηγουμένως, να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας 14. Η κυρία Φερέρα. Ευχαριστώ πολύ. Η, το πρώτο μου ερώτημα είναι περισσότερο σχόλιο. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ε, αυξάναμε τα επιτόκια για να ελέγχουμε τον πληθωρισμό και ο πληθωρισμός ε, συνεχώς αυξάνεται λόγω κερδοσκοπιών στις παγκόσμιες αγορές. Τώρα μειώνουμε τα επιτόκια για να ε, κεντρήσουμε την ανάπτυξη, αυτή όμως δεν έρχεται γιατί υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης στις αγορές και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι πλέον αυτή η σωστή στιγμή να βρούμε τα σωστά εργαλεία και τους σωστούς στόχους μακροπρόθεσμα ή μέσο πρόθεσμα μάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως ε, και το 2010 πρέπει να σκεπτόμεθα ότι θα έχουμε καλύτερη κατάσταση αλλά μην ξεχνάτε ότι το Δεκέμβρη η Κεντρική Τράπεζα προέβλεπε μείωση της ανάπτυξης κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και προχθές Είδαμε τις νέες προβλέψεις για το 2009 που λένε μείωση κατά 1,9% και ε, μείωση της ε, αύξηση με της αναγκαίας κατά πάνω από 9%. Αναφερθήκατε στην συνέντευξή στις 15 Ιανουαρίου και είπατε και παραθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μη συμβατικά μέτρα για να ε, δώσει ανάκαμψη στην οικονομία. Τι εννοείτε με αυτό, μήπως μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, ε, συμφωνώ απόλυτα ε, μαζί σας ότι η εμπιστοσύνη είναι η πεμπτουσία της όλης υπόθεσης αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ε, εμπιστοσύνη στους ιδιωτικούς οργανισμούς, στη συμμετοχή της αγοράς. Έχουμε μία εντυπωσιακή εμπειρία θα έλεγα από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ήμασταν ήδη στην περίοδο των οικονομικών αναταραχών και αυτό το ξέρουμε ε, καλύτερα από τον καθένα γιατί στις 9 Αυγούστου του 2007 τότε ήδη είδαμε ότι θα προκύψουν αναταραχές και τότε θα θυμάστε ε, εφαρμόσαμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις εμπορικές τράπεζες για να διασφαλίσουμε ε, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, 95 δις ε, μετά όμως από αυτή την περίοδο των ε, οικονομικών αταραχών, στα μέσα Σεπτεμβρίου είχαμε ένα γεγονός το οποίο ε, συντενετάραξε συθέμελα την εμπιστοσύνη και στον ιδιωτικό και στον ε, δημόσιο τομέα παντού, στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μοναδικό θα έλεγα και πολύ σημαντικό. Έκτοτε λοιπόν, όπως σας είπα, μειώσαμε ε, τα επιτόκια μας κατά 225 ποσοστιαίες μονάδες, αυτό χωρίς προηγούμενο, με τέτοια ταχύτητα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μείωση των επιτοκίων αυτής της έκτασης, αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ούτε στην Ευρωζώνη και μάλιστα και πριν ε, ε, σαχθεί το ευρώ το 2002. Μιλάμε για μια τεράστια απόφαση η οποία ήθελε να λάβει υπόψη της τις πληθωριστικές πιέσεις, τις απειλές και τους κινδύνους. Σωστά λοιπόν Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της ε, περίοδου είχαμε πληθωριστικές αγωνίες, ε, προσπαθούσαμε να καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα και όσον αφορά αυτές τις ε, πληθωριστικές μας αγωνίες κάπως τα καταφέραμε καλά και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Όπως σας είπα έχουμε μειώσει κατά πολύ τα επιτόκια. Κάτω από το 2% και σχεδόν στο 2%. Βλέπετε λοιπόν τι έχουμε κατά νου. Μέσω πρόθεσμα τώρα, βεβαίω θα θυμάστε ότι το Δεκέμβρη είπαμε ότι ήμασταν στο μείον 1 και στο 0, ήμασταν δηλαδή ε, σε αρνητικό επίπεδο και ήδη τότε αναφέρθηκε ότι πολλοί αισθάνονται ή κίνδυνοι μειώνονται για την ανάπτυξη. Και εγώ ήμουνα σαφής ε, όσον αφορά αυτό εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου το ε, Δεκέμβρη και είπα ότι οι ε, αποφάσεις μας κατά την άποψή μας ήταν αιτιολογημένες γιατί θεωρούσαμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω ύφεση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας που θα ασκούσε περισσότερες πιέσεις. Άρα δηλαδή βλέπετε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την αναζωογόνηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και της πραγματικής οικονομίας. Ανέφερα το γεγονός ότι έχουμε κατά νου να δούμε, σκεπτόμεθα τι θα κάνουμε σε διάρκεια, έτσι ώστε να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, που είναι πολύ δύσκολα. Το γεγονός ότι προσφέρουμε ρευστότητα χωρίς περιορισμό, ε, προφανώς και αυτό δεν είναι στάνταρτ ε, συμπεριφορά μιας κεντρικής τράπεζας. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από την κρίση που βιώνουμε, το να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς χρονικό περιορισμό. Ε, βεβαίως αυξήθηκε κατά πολύ και ο ισολογισμός μας που σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψη μας πάρα πολλές ε, καταστάσεις και εμείς ε, έχουμε εμπλακεί στο να αναλαμβάνουμε κινδύνους σε επίπεδο πολύ περισσότερο από ό,τι συνέβαινε κατά το παρελθόν. Σας τα λέω όλα αυτά για να σας δείξω ότι αυτά που κάναμε κατά το παρελθόν έχοντας πλήρη σεβασμό στην ε, εντολή που μας έχει δοθεί και λαμβάνοντας πλήρη απόλυτα υπόψη τις ε, πληθωριστικές εξελίξεις και την νομισματική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οποτεδήποτε κληθεί είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις και τολμηρές ακόμα. Και ε, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Γκιόμπελς έχει το λόγο. Ε, Τρεις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Μας είπατε και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια της κατά 2,25%. Και αυτό ήταν πράγμα ευπρόσδεκτο. Διαπιστώνουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν βοηθούν τους πελάτες τους, αν θέλετε, να εκμεταλλευτούν αυτή την μείωση των επιτοκίων. Οι εμπορικές τράπεζε εννοώ. Αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους τους και το χρήμα, θέλει θέλετε, περιμένει ακριβό για τους καταναλωτές και ειδικότερα και κυρίως για τις επιχειρήσεις. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνετε δηλαδή και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει η πραγματική οικονομία να αξιοποιήσει την μείωση των επιδοκίων αυτή. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έπαιξε το ρόλο της όπως έπρεπε δηλαδή παρέχοντας ρευστότητα στις εμπορικές τράπεζες. Στην απάντηση, σε απάντηση του κ. Μαργάλιο είπατε ότι διαπιστώνεται μια μικρή ανάκαμψη της διατραπεζικής αγοράς. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Τι σημαίνει ότι οι τράπεζες για δάνεια ενός, δύο μηνών, τριών μηνών, αν θέλετε, παρουσιάζουν, να θέλετε, μια κάποια κάμψη, πτώση. Τουλάχιστον δύο φορές επίσης είπατε, τρίτο ερώτημα αυτό, ότι η οικονομική αυτή κρίση είχε αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι τράπεζες αυτές δεν αποτελούν κομμάτι, τμήμα της πραγματικής οικονομίας, αν θέλετε. Δηλαδή όλα αυτά άπτονται ενός εικονικού κόσμου τελικά. Ή τι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέμπελ. απαντά ο κύριο Τρισέ. Σε ό,τι αφορά την μετάφραση του οποίου στους πραγματικά επιτόκια των σημαντικών ε, μειώσεων στις οποίες προβήκαμε είναι ένα ζήτημα μόνιμο θέλετε και εμείς κινούμεθα με πάσα διαφάνεια. Μειώσαμε το βασικό μας επιτόκιο κατά 2,25%. Και ξέρετε με ποιο επιτόκιο χρηματοδοτούμε τις τράπεζες. Ξέρετε και πολύ καλά μάλιστα. Και καλούμε τις τράπεζες μονίμως και οι εθνικές κυβερνήσεις το κάνουν το ίδιο δηλαδή και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Το σύνολο του ευρωπαϊκού συστήματος θα θέλετε έχει σαφή άποψη από αυτού. Λέμε στο σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών μεταφέρετε αυτές τις μειώσεις με ειλικρινή τρόπο τις μειώσεις των επιτοκίων που εμείς αποφασίζουμε αλλά δεν έχουμε ακόμη πιστεί ότι τα πράγματα όλα γίνονται, όλα που έπρεπε να γίνουν, γίνονται τελικά. Πολλέ φορέ κάποιε από τι παρατηρήσει που γίνονται, θέλετε, είναι αβάσιμε και άλλε φορέ πολύ βάσιμε. Και θα πρέπει να συνεχίζουμε να τι ενθαρρύνουμε και να σπαροτρύνουμε τι τράπεζέ μα. Θα πρέπει να είμαστε όμω προσεκτικοί. Δεν μπορούμε ε, να κατηγορούμε δηλαδή τι τράπεζε ότι στο παρελθόν, θέλετε, αναλάβατε, αν θέλετε, ε, κινδύνου του οποίου ε, ήταν οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα αλλά σε μια οικονομία της αγοράς οι, οι τράπεζες έχουν αυτό ως καθήκον και ως ρόλο δηλαδή. Να κάνουν επιλογή μεταξύ αυτών των κινδύνων δηλαδή. Και εκεί ακριβώς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να είναι εξίσου δραστήριες στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Και αυτό που έκανε η Κεντρική Τράπεζα και αυτό που κάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχει παρά σαν θεμελιώδη στόχο την χρηματοδότηση της ιδίας της οικονομίας μέσω των εμπορικών τραπεζών. Καθήκον και ρόλος των οποίων είναι αυτός εξάλλου. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο σας ερώτημα, τα στοιχεία ανάκαμψης, τα, της προοδευτικής, βραδεία αργής, βραδίας ανάκαμψης της νομισματικής αγοράς, τα βλέπω σε ό,τι αφορά τα επιτόκια τα οποία εφαρμόζονται στην νομισματική αγορά και ειδικότερα τα επιτόκια Euribor ενός μηνός, τριών μηνών, έξι μηνών είπα το επιτόκιο των τριών μηνών που είναι ένα σημαντικό δείκτης για πολλά δάνεια σε ένα μεγάλο αριθμό οικονομιών της Ευρωζώνης. Αυτός θα είναι ο βασικός δείκτης. Αδυνατό να σας πω ότι σε ποσοτικό επίπεδο, σε ποσοτικό καθαρά επίπεδο, έχουμε στοιχεία αρκετά σημαντικά για να μπορούν να θεωρούν, αν θέλετε, ως ουσιώδη. Αυτή είναι μια προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και πάλι εδώ είμαστε, όπως σας έλεγα, επαγρυπνούμε συνεχώς. Τώρα, σημειολογικά να το πάρουμε. Εύκολα μπορεί να είναι κανείς να μιλάει, αν θέλετε, για πραγματική οικονομία και χρηματοοικονομική η πραγματική οικονομία είναι πραγματικά πραγματική οικονομία. Υπεράνω πάση αμφιβολία. Και ω προ αυτό συμμερίζομαι την άποψή σα ότι δεν είναι, αν θέλετε, η κανονική, αν θέλετε, διαχωρισμό που έχει γίνει. Δηλαδή και οι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε και οι καλύτερα από καθέναν στη χώρα σα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τομάτι, αν θέλετε, τη γενικότερη οικονομία. Α μιλάμε λοιπόν για οικονομία και μην κάνουμε τη διάκριση μεταξύ τη πραγματική οικονομία. Κύριε Πρόεδρε, τις ε, τελευταίες ημέρες ε, ακούμε τη μία τραγική είδηση μετά την άλλη από τη Σκοτία, από την Αμερική, ε, απίθανου μεγέθους και διάστασης. Οι κεντρικές ε, τράπεζες με τις υποπτικές αρχές. Είναι εν πάση περιπτώσει θέση να μας πούν ε, κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ή κατά πόσον φτάσαμε στον πάτο. Επίσης, στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν προγράμματα για να αντιμετωπιστούν οι προεκτάσεις της ύφεσης. Έχουμε μείωση του ΦΠΑ στην Βρετανία, φορολογικές ελαφρύνσεις. Δεν βλέπετε να ελοχεύει ο κίνδυνος λόγω αυτών των διαφορετικών ε, προσεγγίσεων του να αυξηθεί η ψαλίδα ε, ανάμεσα ε, στις ευρωπαϊκές τράπεζες και έτσι τα spread για τα κρατικά ομόλογα να διευρυνθούν περαιτέρω αντί να σμικρυνθούν. Τελευταία μου παρατήρηση. Διάφορα ε, νομίσματα έχασαν την αξία τους απέναντι στο ευρώ, κυρίω, η ε, αγγλική λίρα. Όμως ε, η Αγγλία έχει τεράστιο πρόβλημα με τη δική της την κρίση. Αλλά και η Σουηδική κορώνα έχει χάσει κατά 15% από τον Αύγουστο. Και γι' αυτό ερωτώ εσείς ως διοικητής της Κεντρική Τράπεζας πώς ακριβώς εξηγείτε αυτή την εξέλιξη και αυτή η εξέλιξη σα ανησυχεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται ε, μακρηγορώ, σπαταλάω χρόνο στα απαντήσιμο, μου, αλλά εγώ νομίζω οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Από την πρώτη κιόλας μέρα, όταν αποφασίσαμε σε επίπεδο εκτελεστικού συμβουλίου να χορηγούμε ε, δάνεια επί 24 ώρου βάσεως 95 δις ευρώ, τότε πιστεύαμε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική. Και εγώ ποτέ δεν σας είπα ότι βγήκαμε από την δύσκολη αυτή περίοδο. Άρα δηλαδή σας λέω ανεπιφύλακτα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε επί 24 ώρου βάσεως μια καθοριστική στιγμή στη διάρκεια αυτής της επαγρύπνησης ήταν ο Σεπτέμβρης, τα μέσα Σεπτεμβρίου. Γιατί ένα χρόνο μετά την έναρξη των ε, ανατραχών ε, βιώσαμε μια ένταση ε, που απέτησε από εμάς και από αδελφά πιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις μια ειδική απόφαση ειδική παρέμβαση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι, αυτό, ότι ήταν απαραίτητο οι κυβερνήσεις να ε, καταφύγουν σε μέτρα για να ορίσουν μια αμυντική πολιτική απέναντι σε αυτό που εγώ αποκαλώ συστημικό κίνδυνο αφαιρεγγιότητας. Ε, μετά βέβαια αντιμετωπίσαμε και τον ε, κίνδυνο της συστημικής ρευστότητας. Υπάρχει λοιπόν μία άμεση αλληλένδεση ανάμεσα στην οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα που βλέπουμε να εμφανίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Βεβαίως κάτω από αυτές τις συνθήκες εγώ θεωρώ ότι όλοι οι οργανισμοί, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, θα πρέπει ε, να επαγρυπνούν όσο καλύτερα μπορούν για να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, που βεβαίως προϋποθέτουν και σωστή κρίση. Γιατί δεν αρκεί να ε, λάβει κανείς κάποια φορολογικά μέτρα. Αν δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών, το μόνο που καταφέρνει κανείς είναι να επιδεινώνει την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι θα πρέπει να δοθεί όλο το περιθώριο ευελιξίας που υπάρχει στο σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό δεν είναι μόνο ε, μια νομική κίνηση είναι και λόγω συγκεκριμένων παρατηρήσεων που έγιναν στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στο, στις οικονομίες που λέει η αρχή ότι αν χάσει κανείς την εμπιστοσύνη, ό,τι και να κάνει κανείς σε δημοσιονομικό τομέα, αυτομάτως ακυρώνεται από την ε, απώλεια της εμπιστοσύνης. Είναι λοιπόν θέμα αξιολόγησης, ε, σεβασμού του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τον λαμβάνει κανείς υπόψη τους διάφορους ε, οικονομικούς και ε, χρηματοπιστωτικούς ε, περιορισμούς. Δεν θα σχολιάσω το θέμα των κειμενόμενων ισοτιμιών. Βλέπετε υπάρχει κάποια αναταραχή και εκεί, αλλά επανερχόμενος στο πρώτο σας ερώτημα θέλω να πω ότι από τότε που πρωτοεξεκίνησαν οι αναταραχές διαπιστώσαμε ότι το ευρώ λειτουργεί ως ασπίδα για για 300 εκατομμύρια ανθρώπους. Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις. Αντικείμενο, στόχος της Κεντρικής Τράπεζας, πρώτος πρωταρχικός στόχος είναι η εξασφάλιση της ανάπτυξης των τιμών. Κατώτερα αλλά κάτω του 2%. Απομακρυνόμεθα τώρα και από τον στόχο αυτό. Ο αποπληθωρισμός όπως είπατε θα μας οδηγήσει στο 1,5% εκεί περίπου. Μπορούμε να ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί, αλλά παρατηρούμε πως η μείωση του πληθωρισμού από το Σεπτέμβριο είναι υψηλότερη του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και δεν μπορείτε βεβαίως να κατεβείτε κάτω του 0%. Με τη μείωση ΦΠΑ Πιστεύετε ότι θα ε, ε, επιταχυνθεί αυτή η μείωση των τιμών. Γιατί αυτά ακούγονται. Και πώς στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσατε να πείτε ότι θα πρέπει να θέσουμε ένα αμφιβόλο του μηχανισμού αύξηση των μισθών των τιμών. Γιατί οι τιμές μειώνονται. Και δεύτερο ερώτημα, όπως έχουμε κατά επανάληψη πει, τα σχέδια της ανάκαμψης, αναθέρμανσης οικονομιών από πλευράς τραπεζών και αφορά τι τραπέζε δεν οδήγησε σε μια ανάκαψη των υπολείπων τομέων τη οικονομία, μήπω η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική επαναχρηματοδότηση των τιμών στην πραγματική οικονομία μέσω βεβαίω τη Ευρωπαϊκή Τραπέζη Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιπιέτσα. Ο δικό μας ορισμός της σταθερότητας των τιμών είναι λιγότερο από 2% αλλά κοντά στο 2%. Και όταν προηγουμένως μίλησα για την σύνδεση, αν θέλετε, των πληθωριστικών προσοχιών, το είπα αυτό έχοντας κατά νου το λιγότερο 2% αλλά και το κοντά στο 2%. Διότι κατά την περίοδο, κατά τις περιόδους υψηλού πληθωρισμού είχαμε φτάσει στο 4% όπως θα θυμάστε. Αλλά ανέκαθεν αυτό που μας απασχολούσε είναι να είμαστε αξιόπιστοι ότι δηλαδή μπορούμε αν θέλετε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα των τιμών. Και ένα μέτρο για να μπορέσει να μετρήσει τη θέση των τιμών είναι να αναμετρήσει τον πληθωρισμό. Των προσδοκιών δηλαδή, τι οποίε κρατήσαμε στο κάτω από 2%. Κοντά στο 2%. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητώνται αυτή τη στιγμή. Διότι βλέπουμε, αν θέλετε, μια σημαντική αν θέλετε, ελάφρυνση των πληθωριστικών πιέσεων. Αλλά τη στιγμή σα μιλώ αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι έχουμε, αν θέλετε, κάποιε προσδοκίε όσον αφορά τον πληθωρισμό που προσεγγίζουν το 2%. Και ω προ αυτό υπάρχουν σημαντικότερε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Αν δω κάποιου από του δείκτε που λαμβάνουμε εμεί υπόψη, όπου είναι τα index obligations που υπάρχουν, αν θέλετε, κατέρευσαν του Ατλαντικού, γνωστόμαστε πολύ κοντά στις προσδοκίες, αν θέλετε, τον, όσον αφορά τον πληθωρισμό για την επόμενη πενταετία, σε εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή στην οποία βρίσκονται οι ΗΠΑ. Αν συνδέσουμε, αν θέλετε, αυτές τις πληθωριστικές προσδοκίες, σύμφωνα με το δικό μας ονειρισμό σταθερότητας των τιμών, τότε όπως έλεγα προηγουμένως, ο αποπληθωρισμός που παρατηρούμε δηλαδή, είναι καλός δηλαδή. Είναι κατά μία, αν θέλετε, της αγοραστικής ισχύω των οικογενειών και στους οικονομικούς παράγοντες και φορεί εν γέννη. Και αν οι τιμές του πετρελαίου και τη ενέργεια παραμείνουν ε, σε κάποια επίπεδα πολύ χαμηλότερα ευτυχώ και το επαναλαμβάνω αυτό αυτών που έφτασαν στο παρελθόν τότε νομίζω ότι θα έχουμε μια συνέχεια όσον αφορά την μείωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, σε ορισμένα κράτη-μέλη, θα μπορούσαμε μάλιστα να φτάσουμε και σε αρνητικά ποσοστά, τα οποία δεν πρέπει ωστόσο να ερμηνευτούν ως αρνητικά. Αντίθετα, Πρόκειται για μια κατανομή της αγοραστικής ισχύω. Είναι αναπτυξιακό ούτω ή πριν. Και επειδή αυτό όλο συνδέεται με κάποια βασικά φαινόμενα, μέσω πρόθεσμα θα πρέπει να έχουμε έναν πληθωρισμό κάτω του 2%. Κοντά στο 2%, κάτω του 2% πάντω. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ενέργειε και τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα θα έλεγα ότι τάσσομαι αναφανδόν υπέρ αυτών που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εν προκειμένου, επιτρέποντας στις τράπεζες να επαναχρηματοδοτηθούν μέσω και μακροπρόθεσμα προκειμένου να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένας προσανατολισμός ο οποίος συγκρατήθηκε νομίζω επί της αρχής τουλάχιστον από όλους και υπό την παρούσα συγκυρία νομίζω ότι είναι ένας μηχανισμός απολύτως σκόπιμος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γκουε τώρα. Η κυρία Σάρβανεν Μέσου. Η κυρία Βαντερμίς λοιπόν ξεκινάει ή θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η μία ερώτηση έχει σχέση με το πολυσυστημένο θέμα της ε, προφανούς ε, διάστασης ε, ανάμεσα στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των πραγματικών επιτοκίων των τραπεζών. Εσείς είπατε ότι κάνετε έκκληση στο να μειώσουν οι τράπεζες τα επιτόκια, αλλά είναι προφανές ότι αυτές οι εκκλήσεις δεν έχουν καμία επιτυχία. Στη Γερμανία πρόσφατα ακούσαμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα παίρνουν σχεδόν κανένα ε, πλέον δάνειο αλλά και τα επιτόκια είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Ε, δεν πιστεύετε λοιπόν ότι το κράτος ε, το οποίο, το οποίο δίνει δισεκατομμύρια στην αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει το κράτος να έχει λέγει στην διαμόρφωση των επιτοκίων γιατί από ό,τι φαίνεται η αγορά δεν τα κάνει καλά. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά εξελίξεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τις επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. Έχει κανείς εντύπωση ότι αυτή η Federal Reserve, σε αντίθεση με αυτό που είπατε εσείς, ανησυχεί πολύ για τον αποπληθωρισμό. Γιατί αυτό που κάνουν κατ' ουσίαν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί δεν είναι τίποτα άλλο από το να τυπώνουν κατ' ουσίαν χαρτονομίσματα. Ίσως ε, με τον τρόπο αυτό να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να εμποδίσει τον αποπληθωρισμό. Αλλά εκείνο που επίσης είναι σίγουρο είναι ότι τη στιγμή που θα εμφανιστεί η οικονομική ανάκαμψη, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα υπάρξει μια, ένας τεράστιος πληθωρισμός, ε, είναι σχεδόν απόφευκτο. Δεν είναι δυνατόν να τυπώνει κανείς ε, νόμισμα αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή χωρίς κάποια τιμωρία. Τελειώνω. Ε, οι Αμερικανοί ίσως να το κάνουν αυτό σκόπιμα, διότι λόγω της τεράστιας υπερχρέωσης που έχουν, αυτό μπορεί να αποτελεί ένα κομψό τρόπο κάποια στιγμή να ξεκινήσουν από το μηδέν. Εσείς συμφωνείτε με το ότι αυτό είναι μια ηθελημένη στρατηγική και το δεύτερο είναι πώς μπορεί κανείς να αποκόψει την Ευρωζώνη ή είναι δυνατόν και λογικό να αποκόψει κανείς την Ευρωζώνη από όλα αυτά. Τέλειωσα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σας είπα ότι είναι πολύ σημαντικό οι αποφάσεις ε, που λαμβάνουμε να έχετε κατά νου ότι δεν έχουν προηγούμενο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όσον αφορά την έκτασή τους ε η μείωση των επιτοκίων θα έπρεπε καταρχήν να διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία. Συμφωνώ με αυτά που είπατε, είναι πολύ σημαντικά. Και βεβαίως επαναλαμβάνω αυτά που έχω ήδη πει ότι θα πρέπει ε, ο χρηματοπιστωτικός τομέας να λαμβάνει πλήρως υπόψη του αυτά που, αποφασίσαμε. Όμως δεν πρέπει να είμαι απόλυτα αρνητικός. Μιλάμε εδώ για πολλές χώρες όπου οι υποθήκες σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τα τριμηνία επιτόκια του Euribor και υπάρχει σημαντική πτήωση εκεί. Θα έπρεπε λοιπόν ε, αυτό να διοχετεύεται κατά κάποιον τρόπο στα ε, νοικοκυριά σε πολλές χώρες. Εσείς αναφερθήκατε στη στρατηγική εξόδου. Έχετε απόλυτα δίκιο. Οτιδήποτε κάνουμε σήμερα και βεβαίως αυτό ισχύει για όλους μας, για τις κεντρικές τράπεζες, ε, για τα εκτελεστικά όργανα, για το κοινοβούλιο. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνεται έχοντας κατά νου ότι όλα αυτά είναι προσωρινά, είναι στοχευμένα και εμφανίζονται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και πρέπει να έχουμε κατά νου τη στρατηγική οξόδου. Γιατί αλλιώς, όπως και εσείς είπατε, θα είμαστε σε μια ε, συνεχή ε, μεταβλητότητα, ε, μεταπτώσεις, ε, άνοδος και κάμψη και αυτό αν θέλετε είναι η καλύτερη συνταγή για προβλήματα στο μέλλον. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, πρέπει να έχουμε κατά νου. Αυτό που μετράει είναι η μέσο μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Αυτό ισχύει βεβαίω για την Κεντρική Τράπεζα, ισχύει όμως και για τις δημοσιονομικές πολιτικές. Αυτό που χρειαζόμαστε, το πιο σημαντικό κάτω από τις παρούσες συνθήκες, είναι η εμπιστοσύνη και οι πολίτες μας δεν θα νιώθουν εμπιστοσύνη όταν βλέπουν ότι μακροπρόθεσμα ε, δεν έχουμε βιώσιμες στρατηγικές. Η στρατηγική εξόδου από την κρίση είναι καθοριστική σημασίας. να και που μετακυλίονται οι συνέπειες. Οι Ευρωπαίοι σήμερα θέλουν περισσότερη διαφάνεια. Λέτε ότι τους εξωθείτε να μειώσουν τα επιτόκια, όμως τους ρώτησε κανείς ποτέ γιατί δεν το κάνουν. Έχει εξηγηθεί αυτό. Πες ότι αναρωτιούνται γιατί δεν πέφτουν τα επιτόκια. Υπάρχουν λογικές εξηγήσεις αλλά για να κάτσουμε να σκεφτούμε τι μας κάνουν οι τράπεζες Γιατί δεν περνάει η ωφέλη αυτών των μέτρων στους πολίτες, στον κόσμο. Τώρα για την εποπτεία μας είπατε ότι η ομάδα υψηλού επίπεδου εξετάζει πιο μακρόπνες λύσεις. Εσείς προσωπικά όμως πώς το βλέπετε. Μέχρι πού θα πρέπει να φτάσει αυτή η εποπτεία. Τρίτον, ήρθε η ώρα να δοθεί στην τράπεζά σας ισχυρότερη, ευρύτερη εντολή, ούτως ώστε να μπορέσετε να βοηθήσετε την οικονομία της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να έχετε την εντύπωση ότι υποτιμώ τις δυνατότητές μας. για τα επιτόκια και τις συνέπειες για τα νοικοκυριά κλπ. Τα ενυπόθηκα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια, βασίζονται στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Το, το τρίμηνος Λίμπορ, ο τρίμηνος επίσης είναι η βάση του υπολογισμού. Και την Ευρωζώνη και άλλο. Ευτυχώς, οι έχουν πέσει λόγω των αποφάσεων που λάβαμε. Άρα λειτουργήσε το σύστημα αρκετά ενωπητικά. Αλλού τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα. Βέβαια, οι εμπορικέ τράπεζε αντιλαμβάνουν κάποια ρίσκα για να χορηγήσουν τις πιστώσεις και βέβαια θα πρέπει και εμείς να προστατευτούμε έναντι αυτών των κινδύνων. Δεν είναι τα πράγματα απλά, μην τα προστεύουμε. Φυσικά και θέλουμε να υπάρχει όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια. Πάντοτε κάνει καλό. Ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Για την εποπτεία ως ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ε, πρόεδρος της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Έχω να σας πω ότι συμφωνώ με τους πατέρες της Ευρώπης και συνέδρικης του Μάστιχ που προέβλεψαν τη δυνατότητα διεύρυνση της εντολής μας. Στο Δικό Συμβούλιο ανέκαθεν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει όσο γίνεται πιο στενή σχέση μεταξύ Κεντρικής Τράπεζας και Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Και πρέπει πάντα να υπάρχει ε, στεγανό μεταξύ υποπτίας και τράπεζας αυτό ίσως δεν αποδίδει πάντοτε. Δεν είναι τόσο καλή ιδέα. είναι δυνατότητα η συνθήκη, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Έγινε αυτή η επικύρωση εκ των υστέρων. Και τώρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα μια λήψη διαδικασία λήψη αποφάσεων που εμπλέκει και το Κοινοβούλιο. Και είμαστε έτοιμοι για αυτή τη διάβηση τη εντολή. Ακόμα όμω δεν έχει αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, επομένω στην ευρύτερη εντολή, αλλά όχι αλλαγή όσον αφορά την νομισματική πολιτική. Έχουμε την εντολή για μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών που είναι προϋπόθεση για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σας είπα για την πρώτη δεκαετία του ευρώ. Δεν λέμε ότι σήμερα όλα είναι ρόδινα, αλλά γενικά δημιουργήσαν πολύ περισσότερε θέσει εργασία από ό,τι είπα την πρώτη δεκαετία του ευρώ. Euh, euh, euh, Και τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο ερώτα απαντήσεων. Τζον έχετε λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, διερωτώ με κατά πόσον ανησυχείτε για το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίζει να υποβαθμίζει το εθνικό χρέος ε, κρατών μελών και κατά πόσον έχετε κάποια σχέδια έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσετε και την περίπτωση ε, αθέτησης υποχρεώσεων ακόμα και πτώχευσης ορισμένων κρατών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βέβαια δεν είναι φορολογική αρχή. Εσείς έχετε κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ε, στην ομιλία σας ε, σημειώσατε τη σημασία του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είσαστε ευχαριστημένος με το ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πλέον ε, θα μπορούσε να καταρτήσει κάποια σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αναφερθήκατε στις ισοτιμίες ε, στην ομιλή σας, αλλά μήπως πιστεύετε ότι το όλο θέμα πρέπει λιγάκι να το επανεξετάσει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα ακριβώς αυτό που θέλετε να πείτε με τις ισοτιμίες. Δηλαδή εσείς είσαστε κατά ε, των ισοτιμιών και θέλετε να υπάρχει σταθερότητα των τιμών όσον αφορά το ευρώ. Αλλά υπάρχουν άλλα ε, νομίσματα ε, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην Ευρωζώνη. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας συντονισμός έτσι ώστε να έχουμε και σταθεροποίηση των νομισματικών ισοτιμιών. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, Γνωρίζετε ότι η θέση μας ανέκαθεν ήταν ε, ξεκάθαρη. Οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνε για τη φορολογική τους πολιτική. Πρέπει να παραμείνουν επιστές ε, στο σύμφωνο σταθερότητας και θα θυμάστε ότι παλαιότερα είχαμε τεράστιες πιέσεις για να ακυρωθεί το πρόγραμμα αυτό. Όχι βέβαια από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν συμφωνούσε. Και πρέπει να σας πω ότι και εμείς οι ίδιοι λέμε ότι βρισκόμαστε ε, σε μια περιοχή ενιαίων νομίσματος, ε, το σύμφωνο σταθερότητας ε, είναι κατ' ουσίαν η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Άρα δηλαδή οι κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσει. Και ήδη είπα ότι το σύμφωνο σταθερότητα δεν ε, επιβάλλει απαραίτητα τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούμε, αλλά είναι ένα σημείο αναφοράς, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Γι' αυτό λοιπόν ε, παραμένω σε αυτό και υπολογίζω και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να ασκήσουν έλεγχο πιστικά. Δηλαδή δεν ανησυχώ ιδιαίτερα, ήδη ανέφερα ότι η ιδέα να αμφισβητηθεί το ευρώ ή η ευρωζώνη, αυτό για μένα είναι εκτός θέματος που όπως σας είπα και πάλι είναι οι κυβερνήσεις να επανέλθουν σε μια περισσότερο βιώσιμη πολιτική. Αυτό είναι ένα ε, θέμα που συζητιέται επανειλημμένα. Όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είπα με απόλυτη σαφήνεια ότι κατά την άποψή μου η εντολή επιτήρησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να προβληθεί περισσότερο γιατί χρειαζόμαστε απαραίτητα ένα ισχυρό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, συμφωνώ με αυτά που λέχθησαν όχι όμως για την Ευρώπη και σίγουρα όχι για την Ευρωζώνη, γενικότερα για τον κόσμο ότι είναι απαραίτητο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει καταστάσεις που είναι δύσκολες και ε, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, εκεί νομίζω ότι το Διεθνές Ζωμανιστικό Ταμείο είναι ιδιαίτερα ενεργό. Όσον αφορά την πολιτική σου δεν έχω τίποτα να προσθέσω επ' αυτού. Υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν και άλλα που δεν αλλάζουν. Ο κύριος Λάου και ο κύριος Χινάς καταρχήν. Κύριο Λάου καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κύριε Τρισέ τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η μία κατ' ουσίαν ετέθη ήδη η διαφορά spread ε, μεταξύ Ελλάδας, ε, Ιρλανδίας, ε, Γερμανίας και άλλων χωρών διευρύνεται στην Ευρωζώνη. Θεωρείτε ότι αυτό είναι πρόβλημα για την Ευρωζώνη και πόσο μπορεί να αντέξει η Ευρωζώνη. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για τα επισφαλή δάνεια. Θεωρείτε ότι αυτό είναι πρόβλημα ή να το πω αλλιώς Πώς, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διαρθρωθεί μια τράπεζα. Τώρα τα παράγωγα. Αν καταρρεύσει η αγορά των παραγόγων, νομίζω δεν θα υπάρχει σωτηρία. Εσείς βλέπετε αυτή τη στιγμή να υπάρχει πρόβλημα ε, αθέτησης υποχρεώσεων από πλευράς της αγοράς των παραγόγων. Και Όσον αφορά τα ε, παράγωγα, υπάρχει ανοιχτή ανταλλαγή ή υπάρχει κάποια επιτήρηση. Ε, Για την ε, διαφοροποίηση που επικρατεί στην Ευρωζώνη. Από την αρχή λοιπόν ακούγονταν και ακούγονται αυτές οι παρατηρήσει. Διαφορετική ρυθμή ανάπτυξης, διαφορετική δείκτες πληθωρισμού, διαφορετική εξέλιξη των ε, δικτών. Εμείς το προσεγγίζουμε ιδιαίτερα προσεκτικά και το προσεγγίσαμε από την αρχή και κάναμε και συγκρίσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι κάτι το ασύνηθες δηλαδή να υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα, αυτή η διαφοροποίηση. Παρατηρούμε δε ότι η τυπική απόκληση της ανάπτυξης του πληθωρισμού επίσης, του πληθωρισμού, οι διαφορές ε, που υπάρχουν δηλαδή δεν είναι διαφορετικές οι ΗΠΑ από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από πολιτεία σε πολιτεία στην, ε, στην Αμερική και από κράτος σε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς μιλούμε δηλαδή για την φορολογική κατάσταση μιας σειράς κρατών μέλων. Θα έλεγα ότι σε όλα τα κράτη-μέλη πλέον υπάρχει αυτή η δυσκολία και γι' αυτό λοιπόν είπα ότι η στρατηγική εξόδου είναι σημαντική για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Εσεί μιλήσετε για τέσσερα μόνο κράτη-μέλη, αλλά και για τα δύο που έχουμε εμεί κατά νου. Αν θέλετε, που έχουν καλή συμπεριφορά, η, η στρατηγική εξόδου δηλαδή είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αλλά είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να η εκτελεστική κλάδη και τα κοινοβούλια δηλαδή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αναλογιστούν τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν. αλλά είναι ένα επιπλέον ισχυρό επιχείρημα και το λέμε αυτό ευθύ εξ αρχή, από την πρώτη στιγμή δηλαδή. Λέμε ότι έχετε αυτή την ευθύνη. Εσείς θα πρέπει να συμπεριφερθείτε. Και το Σύμφωνο Ανάπτυξης σταθερότητα δεν είναι ένα έτσι αφαιρημένο πλαίσιο. Που θα θυμάστε ότι τριών ετών, τεσσάρων ετών ακούστηκαν αυτά. Ότι είναι κάτι το αφηρημένο, είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο αυτό του Συμφώνου Ανάπτυξης Σταθερότητας αν θέλετε, και ότι θα πρέπει να βασίζεται και να εδράζεται, αν θέλετε, σε πολύ ισχυρά οικονομικά στοιχεία. Η πίεση όμως ε, της συγκυρίας και της πραγματικότητας θα ελπίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν το θεωρώ δηλαδή αυτό ότι αυτή η έννοια θέλετε αυτής της ανεύθυνης, ας την πούμε έτσι, κακής τράπεζας ισχύει και όσο ό,τι αφορά τον κλάδο και τον τομέα των παραγόγων, όπου είχαμε μια έκρηξη, αν θέλετε, των ε, θεωρητικών ποσών για όλα, αν θέλετε, τα παράγωγα και ειδικότερα για τα credit default swaps πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε επίγνωση γεγονότο ότι υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, ο οποίο έχει ήδη εντοπιστεί και έχει αναγνωριστεί, και το λέω αυτό τακτικά, όπω επίση και σε όλε αυτέ τι επισκοπήσει που γίνεται τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωπαϊκής. Θα πρέπει να στηριχθούν, αν θέλετε, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι κεντρικοί μας ομόλοι, οι τράπεζες δηλαδή. Είναι ένα σημαντικό βέβαιο που συνοθεί κατεύθυνση και το οποίο υποστηρίζουμε. Ο κύριος Σινάς. Τον κάνουμε αυτό τώρα. Θα διαπιστώσετε πρόσφατα ότι κυκλοφορούν ευθύμες, εικασίες γίνονται και κριτικές από τους ευρωσκεπτικιστές ειδικότερα που επιτίθενται στο ευρώ στοχεύοντας να θέλετε τα spread και το πράττουν αυτό κατά τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία όσον αφορά τις πραγματικές προθέσεις. Οι πραγματικές προθέσεις θα θέλετε είναι το ευρώ το ίδιο. Και εστιάζουν σε αυτόν. Χθες η Ελλάδα υπέστη αυτή την επίθεση και ο κύριος Αλμούνιο Επίτροπος ήταν κατηγορηματικός απαντώντας σε ένα ερώτημα της Προέδρου είπε ότι όλοι στο ίδιο καράβι, στην ίδια βάρκα βρισκόμαστε. Είπε ότι έχω την εμπιστοσύνη μου, δεν ανησυχώ, είπε ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, αλλά στην Ευρωζώνη δεν τίθεται ζήτημα αν θέλετε προσφυγής, αν θέλετε σε εξωτερικά μέσα, σε διεθνεί άλλους οργανισμούς. Και είπε ότι δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να απαντήσουμε δηλαδή σε εκείνους που ποτέ δεν θέλησαν το ευρώ και σε εκείνους αν θέλετε τις ε, υπηρεσίες αξιολόγηση που είδαν το παγόβουνο να προσεγγίζει, να πλησιάζει, αν θέλετε, ε, το παγόβουνο να πλησιάζει το Ιδανικό και τώρα ανακαλύπτουν, δεν έκανα τίποτα και τώρα ανακαλύπτουν ότι η Ισπανία, η Ελλάδα δηλαδή, αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες Θα ήθελα δηλαδή με τον ΑΒ τρόπο, βεβαίως εσείς απαντήσατε, θα ήθελα, αν θέλετε, να μου δώσετε αυτή την ε, πιο στοχευμένη, αν θα μπορούσα να την αποκαλέσω έτσι, επιβεβαίωση. Ευχαριστώ. Επιβεβαιώνω απολύτω αυτά τα οποία είπα. Και έχω πει σχετικά με τη χώρα σας, αλλά και άλλα κράτη-μέλη ενδεχομένω θα έλεγα, ότι η ευθύνη έγκυται και βρίσκεται στην Αθήνα. Θα πρέπει η Αθήνα να διεξάγει, αν θέλετε, βιώσιμες αιφόρε πολιτικές μακροπρόθεσμα και πιστικές συνάμω σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, επίσης όμως και στο επίπεδο, αν θέλετε, της σχετικής ανταγωνιστικότητας των μοναδιών κόστους παραγωγής, που είναι πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το μήνυμα, το συνεχές, το διαρκές μήνυμα που ήδη εμείς απευθύνουμε στο σύνολο των κρατών της Ευρωζώνης αδιακρίτως. Αδιακρίτως, χωρίς καμία διάκριση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η σταθερότητα της Ευρωζώνης δεν αμφισβητείται. Αν το ευρώ δεν ήταν στέρεο, αυτό θα φαινόταν. Κανεί δεν το αμφισβητεί αυτό. Όλα τα νομίσματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση που είναι μια κατάσταση προφανώ πραγματικών δυσκολιών. Αυτό είναι αδιασφυσβήτητο και εμφανέστατο, πρόδειλο. Αυτό ισχύει για όλα τα νομίσματα του κόσμου τα οποία προσωπικώ γνωρίζω και δεν θα ανακατονομάσω κάποιο συγκεκριμένα, αλλά όλοι θα αναγνωριστείτε ούτω ή Α σταθείτε δηλαδή στο ύψο των ευθυνών σα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο συνεχώ και, και διαρκώ προσπαθούμε να περάσουμε. Για τη συλλογική ομάδα, η κυρία Βανερμπόρτ τώρα. Yeah, thank you. Um, Ευχαριστώ. Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα ε, όλο αυτό το μήνυμα το οποίο στείλατε για την εποπτεία και θεωρώ πολύ θετικό το ότι τώρα στην Κεντρική Τράπεζα υπάρχει προβληματισμός σε σχέση με την εντολή της. Διαφωνώ για το FSF ελαφρώς σε σχέση με το ποιοι φορείς εκεί συναντώνται γιατί κατά τη γνώμη μου πρόκειται μόνο για ένα τμήμα του τραπεζικού κόσμου. Άλλωστε, οι ρίζες της κρίσης βρίσκονται εκτός του τραπεζικού τομέα. παράγοντα, είπατε, τα OTC. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και κάποιους εμπειρογνώμενες από τα χρηματιστήρια και να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό όπως και στο παγκόσμιο σύστημα εποπτείας. Άρα, τι λέτε, ε, εσείς στην Κεντρική Τράπεζα ε, θέλετε να είστε ένα τμήμα αυτού του γενικού του συστήματος ή να έχετε αυτόνομο ρόλο. Σας ευχαριστώ, λίγο Όχι, όχι. Δεν ξέχασα αυτό το οποίο προτείνατε. να πω ένα μήνα. Πάντα το έχουμε υπόψη μας. Τώρα όσον αφορά το FSF, δεν είναι μόνο αυτό το άτυπο βήμα της ε, Επιτροπής της Βασιλείας. Άλλωστε ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας εκεί προεδρεύει. Εκεί συναντιούνται λοιπόν επιτροπές χρηματιστηρίων, η Παγκόσμια Τράπεζα, ε, κεντρικές τράπεζες. Ε, επομένως πρόκειται για αυτό το άτυπο φόρουμ. Ε, γι' αυτό λέω ότι εκεί συναντώνται όλοι όσοι εμπλέκονται στο τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίω και το ρίζο του κακού δεν είναι το τραπεζικό σύστημα. Κάθε άλλο. Είναι όλοι όλοι όμω εκεί. Και μπορεί να βελτιωθεί άμα γίνει ακόμα ευρύτερο. Έχουμε επομένω εκεί πέρα και εκπρόσωποι τη εξουσία και ανεξάρτητου φορείς ανεξάρτητου από την πολιτική όπω η, η Επιτροπή τη Βασιλείας, άλλε συναφείς επιτροπέ και οι Κεντρική Τράπεζα. άτυπο λοιπόν βήμα, άτυπο, άτυπο φορέας είναι όπου όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες μπορούν να βρουν τη σωστή πορεία και μετά βέβαια εξαρτάται από την σοφία του να βρεθεί λύση. Κυρία Φαντερμπερκ, θέλετε να δευτερολογήσετε. Ναι, ναι. Κυρίως στο ότι ε, από μόνοι τους κεντρικοί τραπεζίτες δεν μπορούν να καλύψουν όλο αυτό το φάσμα των θεμάτων. Γι' αυτό και χρειάζεται να το συζητούμε εδώ στην Ευρώπη για τα χρηματιστήρια, για όλα αυτά, όλα όσα έγιναν. Έχετε δίκιο, αλλά οι κεντρικές τράπεζες ε, παρόλα αυτά ε, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι μοναδικές ε, με την έννοια ότι δεν έχουν δικά τους συμφέροντα από το Σύνταγμα έχουν αναλάβει το να έχουν κατά νου τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και αυτό τη καθιστά μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να πω ότι αν δούμε όλους τους θεσμούς που υπάρχουν στον κόσμο, αυτοί οι θεσμοί που είναι πιο ξεκάθαροι είναι ε, η BIS και οι ίδιες οι κεντρικές ε, τράπεζες ε, είναι δηλαδή μοναδικές ε, στο να προσφέρουν την μέσο μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Σας τρεις ερωτήσεις. Ο Πόμος μας είπε για τις ισοτιμίες και δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω. Όμως υπάρχει μια πρώτη συμφωνία όσον αφορά την νομισματική συμφωνία. Τίποτε θα γίνει όσον αφορά την διεθνή αρχιτεκτονική. Αυτό είναι άσχετο με το τραπεζοπιστωτικό σύστημα. Και με τον αναδυόμενο προστατευτισμό. Κάτι άλλο θα, ήθελα να μας πείτε. Τι λέτε για την παγκόσμια οικονομία, γιατί αυτή η κρίση χτύπησε περισσότερο τους στοχούς. Οι αναδυόμενες οικονομίες, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες χτυπήθηκαν πολύ περισσότερο. Επομένως, θα έπρεπε αυτόν έχουμε κατά νου όταν θέλουμε να ξανασχεδιάσουν το σύστημα. Δεν αρκεί ούτε το G20 ούτε το FSF. Χρειάζεται ένα G92, ξέρω Επίσης, αυτό έχουμε το πρόβλημα με την ρευστότητα μεταξύ ενεργητικού και παθητικού που είναι το, είναι το σημείο ισορροπίας. Γιατί να έχουν τόσο περισσότερο περιθώριο τα τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα τα αμερικανικά από τα δικά μας. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη ερώτηση. Ήδη σας είπα δεν έχω τίποτα να σας πω ιδιαίτερα όσον αφορά τις ισοτιμίες απλώς. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σας αναφέρω το ότι αυτό στο G7 στα κειμενόμενα νομίσματα το συζητήσαμε και ξέρετε καλύτερα από όλους όλους ότι οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις ασχοληθούν πάρα πολύ με το θέμα. Και έμειναμε σταθεροί σε αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στις αναδειόμενες οικονομίες. Και κυρίως για την Κίνα το είπαμε. Τα είπαμε και γι' αυτό μην περιμένετε να διαφοροποιηθώ σε σχέση με τα συμπεράσματα του G7. Τώρα όσον αφορά για το πρόβλημα της φτώχειας και την παγκόσμια οικονομία συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες χωρίς να έχουν ενεργειακή παραγωγή, χωρίς ε, εμπορεύματα, αυτά τα οποία ευνοεί η παγκόσμια οικονομία, αυτές οι οικονομίες, αυτά τα κράτη βρέθηκαν στη χειρότερη θέση. Η δε πτώση της τιμής των ε, καυσίμων κάπως, κάπως, κάπως διευκόλυνε τα πράγματα για αυτές τις χώρες. μέσα σε αυτό το κλίμα της υπερβαινόμενης οικονομίας. Όχι, το, το G20 δεν είναι η παγκόσμια οικονομία. Είναι όμως ένα φόρουμ άτυπο εκεί που είναι δυνατόν να διαμορφωθεί συνένεση για ένα σωρό σημαντικά ζητήματα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο μετά την κρίση στην Ασία και τώρα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σημαντικό ακριβώς αυτή την πορεία προς το να οριμάσει ένα συμβασμό, μια συνέντευξη. Α πούμε κάτι για του Διεθνές Ταμείο ότι διαμορφώνεται και ένα κλίμα και το οποίο μετά πηγαίνει προ συζήτηση η προβληματική αυτή στο διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, έτσι δουλεύει το σύστημα. Πολύ σημαντικό αυτό που ρωτήσατε και τώρα για το τι κάνουμε εμείς. ήταν η πρώτη κεντρική τράπεζα στον κόσμο που δεσμεύθηκε με, αυτό το, το, αυτή την τριμηνία και εξαμηνία αναχρηματοδότηση. Κανείς πριν την κρίση δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο όμως. Υπάρχουν κάποιες ε, εξαιρετικές πράξεις αγοράς ε, χαρτοφυλακίων τις οποίες προβαίνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον είπα, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε τέτοια κίνηση. Μπάς περιπτώσει όμως επαγρυπνούμε συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, για πάρα πολλά χρόνια ήσασταν υπέρ των ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε αποτελεσματικούς τομείς της οικονομίας. Τώρα έχουμε ένα τομέα που ήταν αποτελεσματικός, τώρα όμως σημειώνει μεγάλη ζημιά. Είναι ο τραπεζικός τομέας. Έχετε κατά νου να εφαρμόσετε διαρθρωτικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη η ομάδα του κυρίου Walker ε, κατέβαλε προτάσεις ε, σχετικά με τη λιανική, τραπεζική ε, και πολλές άλλες προτάσεις σχετικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα. Θεωρείτε ότι και εδώ στην Ευρώπη μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους προτάσεις. Όπως σας είπα, πρέπει να μην επιδεικνύουμε αυταρέσκεια οποτεδήποτε σχολιάζουμε το, τα οικονομικά συστήματα. Η λειτουργία της ε, αγοράς έτσι και αλλιώ από μόνη της ε, θα προκαλέσει αναδιάρθρωση και αναμόρφωση της βιομηχανίας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να βοηθήσουμε στην σωστή αναδιάρθρωση και αναμόρφωση να ακολουθεί σωστή κατεύθυνση, πολύ σωστά είπατε ότι ο τομέας αυτός ε, πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Οφείλουμε λοιπόν να τροποποιήσουμε, να βελτιώσουμε τους ε, κανονισμούς. Ε, εγώ δεν έχω ακόμα τη δυνατότητα εκ μέρου ε, του Διοικητικού Συμβουλίου να σχολιάσω αυτή την έκθεση, αλλά την εξετάζουμε πολύ προσεκτικά και πρέπει να πω ότι αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες αυτό ήταν ε, περισσότερο αμερικανικό προϊόν και ξέρετε ε, για μας επειδή δεν υπήρξαν συγκεκριμένες αποφάσεις τελικά αποδείχθηκε άχρηστη αυτή, αυτός ο διαχωρισμός, άχρηστος. Στην Ευρώπη έχουμε μια διαφορετική έννοια τραπεζικών συναλλαγών. Δεν υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα σε επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες. Έχουμε ε, γενικών δραστηριοτήτων τράπεζες. Οι τράπεζες ασχολούνται και με επενδύσεις ε, και με εμπορικές συναλλαγές και με λιανική τραπεζική. Αυτό ίσως είναι και καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο κρίνοντας και από τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς ε, θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε όλα αυτά πολύ προσεκτικά. Όπως σας λέω αυτά είναι σκέψεις ε, παγκοσμίου κλίμακας. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα τολμηρό τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομίες της αγοράς δεν είναι τόσο τροτές και έχουν και την δυνατότητα απορρόφησης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ε, ξαναεμφανιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι τώρα μία δοκιμή αυτή που γίνεται και ε, πρέπει να βρούμε ε, τις λύσεις για το μέλλον. Να έχουμε αμορτισέρ, προφυλακτήρες στην παγκόσμια οικονομία, αναχώματα για να είμαστε πολύ πιο ανθεκτικοί. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στις τέσσερις τελευταίες ερωτήσεις για το ΕΛΚ. Ο κύριος Πέτσακ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση προθέρμανσης. Ποια είναι η πρώτη αξιολόγηση όσον αφορά την προσχώρηση, την ένταξη της Σλοβακίας στην Ευρωζώνη και ποια θα είναι ο αντίκτυπος στις τέσσερι ελευθερίες εσωτερική αγοράς. Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων καταρχήν και την οδηγία για τις υπηρεσίε, Τι θα γίνει. Αν θα έχει θετικό αντίκτυπο. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξή: Πώς βλέπετε, πώς πιστεύετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορέσει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη στα προβλήματα ρευστότητος που αντιμετωπίζουν και στην περίπτωση αυτής της κρίσεως με διαφορετικές συμφωνίες που είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται αυτή τη στιγμή σε περίπτωση κρίσεως θα μπορούσε αυτό να περιορίσει την ροή κεφαλαίων, δηλαδή μεταξύ των ε, κεντρικών και των ε, θηγατρικών τραπεζών και στα κάτι μελη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πώς πιστεύετε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δώσει λύση στα προβλήματα πληρωμών που αντιμετωπίζουν και στο Το ότι ο, ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο Ντομινίκ Στροσκάν, να πούμε, εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τη Σλοβακία, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι έγινε, έφτασε αρκετά καλά, θα έλεγα. Διαπιστώσαμε ότι από τεχνικές απόψεις υπήρχε τέλεια προετοιμασία, άψογη προετοιμασία και τις προφορίες τις οποίες εισέλαβα τόπου δηλαδή, γιατί και εμείς συμμετείχαμε ενεργά σε αυτή την ε, αλλαγή δηλαδή, όλα τα στοιχεία, οι δείκτες είναι ενθαρρυντικοί και βίωνοι. Και πιστεύω ότι η Σλοβακία θα ενταχθεί επιτυχώς στην Ευρωζώνη. Και 10 χρόνια μετά το ευρώ βλέπουμε ότι πλέον 16 είναι τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν ε, στην ε, Ευρωζώνη μαζί με τη Σλοβακία. Το πλέον πρόσφατο μέλος αυτής. Όπως γνωρίζετε, Έχουμε σχέσεις με τα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων και τη δική σα τη χώρα, τη Σλοβακία δηλαδή, και δεν θα επεκταθώ άλλο. Χρήσιμο είναι που βρέθηκε ο τρόπο βεβαίω να στενή συνεργασία ε, με την Κεντρική Τράπεζα τελικά και σε άλλε περιπτώσει δεν χρειάστηκε, δεν στάθηκε αυτό απαραίτητο, αλλά συνεχίζουμε τις επαφές μας και τις στενές μας σχέσεις με όλε τι κεντρικέ τράπεζε των 100 μελών τη Ευρωπαϊκή Ενώσης Και σε ό,τι αφορά το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, σημειώνω αυτά που είπατε. Σε ορισμένε περιπτώσει που θα γνωρίζετε, η παρουσία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου θεωρείται χρήσιμη από την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση τη οικία χώρα. Ο Πίτροπος Σαλμούνια νομίζω σας είπε ότι μπορούσε να σας πει όσον αφορά τη συμβολή και τη συνεισφορά του διεθνού της Ευρωπαϊκής Ενώσεω μέσω αυτής της διευκόλυνσης του facility που θα μπορούσαν να εργοποιήσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που αποτελεί και αυτή μια σημαντική συνεισφορά και συμβολή δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει τις παρατηρήσεις σας τις σημείωσα. Η ε, κυρία Λούλινγκ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε κατά τρόπο μεμονωμένο θα έλεγα έναν μεγάλο αριθμό οδηγιών για την ε, δομή και την αρχιτεκτονική της εποπτείας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που θα μπορούσε να κατηγορηθεί για όλα τα δεινά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να μας βγάλει από αυτή την κρίση. Καλούμεθα να λάβουμε συγκυριακά αποφάσεις, περιστασιακά αποφάσεις, ώστε να ξέρουμε Πού πηγαίνουμε. Αν θέλετε είμαστε σαν τεχνίτες που εργάζονται, αν θέλετε, χωρίς αρχιτέκτονα και χωρίς την επίβλεψη και την εποπτεία. Και βλέπετε και φαντάζεστε τελικό, το τελικό οικοδόμημα σε τι κατάσταση θα μπορούσε να καταλήξει. Κάποια θεσμικά όργανα βεβαίως μέσα σε αυτή την περίοδο κρίσεως, μεσούσε τη κρίσεω δηλαδή, κινήθηκαν και πορεύτηκαν προς την ευρωπαϊκή αλλά λιγότερο. Πιστεύετε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να αναγκαστεί να διευρύνει το πεδίο αρμοδιοτήτων τη ειδικότερα και κυρίω σε ό,τι φορά την εποπτεία, διότι πολλέ, αν θέλετε, φωνέ ακούγονται υπέρ και πιο συγκεκριμένα και τι θα γίνει δηλαδή με τις χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης. Και το τελικό με ερώτημα. Θα θέλατε κι εσείς ε, να ασχοληθείτε με αυτούς τους ε, εταιρείε και τους οργανισμούς, να θέλετε αξιολόγηση του ελληνικού εικονότητος, γιατί όπως έχει αυτή η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι σχετικά μπλεγμένη. Ο κύριος Τρισέ, σημειώνω βεβαίως την, ε, και, την περιπλοκότητα της καταστάσεως και τις παρατηρήσεις ε, σας όσον αφορά τις ε, δυσκολίες να βλέπετε δηλαδή εργάτες να κάνουν τη δουλειά τους αν θέλετε με τον πιο ευσυνείδητο τρόπο και ενσυνείδητο τρόπο αν θέλετε χωρίς να διαθέτουν αρχιτεκτονικά σχέδια. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καρό παράδειγμα θέλετε. Σας είπα πού βρισκόμαστε ποιες είναι οι δικές μας σκέψεις, ποιες είναι οι δικές σας ε, σκέψεις, εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή και της ομάδος ε, υπό τον κύριο Ντεβαροζιέρ και εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε και να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απευθύνονται. Σαφώς υπάρχει ένα διέξοδο που έχει ήδη προαποφασιστεί θα έλεγα και κατά κάποιο τρόπο από εκείνους που συνέταξαν τη συνθήκη του Μάστρικτ και που κυρώθηκε από το σύνολο των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων ε, δημοψηφίσματος δηλαδή και εμείς ενεργούμε πάντα υπέρ μια στενή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ε, αρχών τραπεζικής εποπτείας των κρατών μελών. Τώρα για τους αυτούς τους εταιρείε αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητος. Έχουμε ήδη αρκετές ευθύνε. Ίσως να αναλάβουμε και άλλες νέες ευθύνε. Πρόκειται πάντως για ένα μείζον ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζουμε, γιατί πρόκειται για ένα από τα σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικότατα. Είναι σαφές αυτό. Και είναι ένα σημείο για το οποίο επιμένω θα πρέπει να υπάρξει διατλαντική συμφωνία. Διότι βρισκόμαστε στο πλαίσιο ενός παγκοσμιωμένου συστήματος και είναι απαραίτητο να βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα αυτό που με με κατέρωθεν του Ατλαντικού. Πρόκειται πάντως για ένα πολύ μείζον θέμα το οποίο ε, θέσατε. Κύριε Πρόεδρε, να σας θέσω και εγώ κάποιε ερωτήσει θα ήθελα, γιατί συμμερίζομαι με την κυρία Λούνη την ιδέα ότι εργαζόμαστε χωρίς αρχιτέκτονα, χωρίς μηχανικό δηλαδή. Γι' αυτό και απορρίψαμε μια πρόταση που έγινε όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση που έγινε. Αλλά έχουμε την οδηγία για την κεφαλιακή επάρκεια και θα θέλαμε τη γνώμη τη Κεντρική Τράπεζα, την οποία ελπίζουμε να λάβουμε. Και εγώ έχω αυτή την εντύπωση, εργαζόμαστε χωρί μηχανικό. Αν θέλετε και με τρόπο, αν θέλετε, παλαιωμένο, απερχαιωμένο. Γιατί μα είπαν ότι η αναθεώρηση τη επανεξέταση αυτή τη οδηγία κεφαλαίου και πρέπει να γίνει για να ληφθεί υπόψη του off-balance sheet, προβλήματα εποπτεία, προβλήματα ρευστότητο ξέρω και ενδεχομένω ίσω να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, και προβλήματα ιδέε. Όπω επίση και να απαιτήσεων για τα hedge funds. Γιατί όχι, αν θέλουμε να υιοθετήσουμε μια πιο υφή προσέγγιση στι χρηματαγορέ. Τι πιστεύετε για αυτή την νομοθετική πρόταση η οποία μα έχει και την οποία εξετάζουμε και έχουμε δεσμευτεί να λάβουμε θέση πρώτου τέλου τη θητεία μα. Όσον αφορά τώρα το G20, συμμερίζεσαι εσείς την προσέγγιση και την άποψη σύμφωνα με την οποία αυτά που έγιναν το τελευταίο τρίμηνο ήταν πολύ καλά, εκτός όμως ό,τι αφορά το μακροοικονομικό σκέλος θα μπορούσαμε να κάνει κάτι παραπάνω. Αναφερθήκατε επίσης στα προβλήματα τα σχετικά με την εποπτεία. Αν βγούμε, αν εξέλθουμε αυτή την κρίση χωρίς να έχουμε αντιμετωπίσει τα, τη ρίζα και τι τις οικονομικές αν θέλετε παγκόσμιε ανισορροπίες δεν θα έχουμε πολύ προοδεύσει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν σχέδια αναθέρμανσης αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα της παγκόσμιας αστυνομίας που βρέθηκε, αν θέλετε, στην απαρχή αυτών των εκτροπών που διαπιστώθηκαν και παρατηρήθησαν στις χρηματαγορές. Συμμερίζετε την άποψη αυτή. Πείτε μου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε ενεργότατα και δραστήρια στην επεξεργασία της γνωμοδότησής μας ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις κεφαλικές απαιτήσει και θα τη λάβετε συντομότατα. Ευχαριστώ την προσοχή σα σε ένα σημείο. Ότι μα αν θέλετε, αν θέλετε, στο πλαίσιο αν θέλετε, μιας παγκόσμιας συζήτησης που γίνεται όσον αφορά το πρακτέο δηλαδή για να μπορέσουμε να διδαχθούμε και να αξιοποιήσουμε τα διδάγματά μας στο πλαίσιο αν θέλετε της, ε, το financial stability και στο πλαίσιο της βασιλείας εργαζόμαστε σκληρά προς την κατεύθυνση αυτή. Και όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να διαχειριστεί, αν θέλετε, το, να διαχειριστούμε μάλλον το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, διότι διαφορετικά όλοι βρισκόμαστε στο έλεος, αν θέλετε, μιας έκρηξης η οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί εδώ ή εκεί. Η οδηγία αυτή έρχεται μάλιστα σε μια στιγμή που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν θα πρέπει να κάνουμε τα λάθη αντλώντας τα διδάγματα δηλαδή από την κατάσταση αυτή που προηγήθηκε. Γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί, αν θέλετε, να τα ξαναδούμε όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό ισχύει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Παντού δηλαδή. Η παγκοσμιοποίηση του συστήματος, του οικονομικού συστήματος, του χρηματοοικονομικού συστήματος, του διεθνούς, σε όλους μας δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής και επιμονή μου βάσος θα έλεγα διαρκώς για το G20. Συμμερίζομαι απολύτως στα συναισθήματά σα και την άποψή σα. Για μια ακόμη φορά όμω και όπω σα είπα προηγουμένω. Ο θεσμό δει ούτως πριν για να μπορέσει να ασκήσει εποπτεία αν θέλετε. Με πραγματική ικανότητα να αλλάξει τα πράγματα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο ασκεί, αν θέλετε, αυτή τη μακροοικονομική και μακροοικονομική εποπτεία με θέση ανανεωμένη θα έλεγα, ανανεωμένη εξουσία θα το πούμε έτσι. Διότι αν όλα θα μας οδηγήσουν στο status quo άντε, με το ίδιο έλλειμμα Φερρυπίν και τις ανισορροπίες αυτές, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές, τότε θα βρεθούμε ακριβώς στην ίδια θέση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Και δυστυχώς, και δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε και ενδεχομένως και νέα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε σημαντικά την εποπτεία, την μακροοικονομική εποπτεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να το πετύχει αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Η κυρία Μπαϊδά. Ευχαριστώ ah, κυρία Πρόεδρε. αν κάτσουμε να υπολογίσουμε πως είναι σήμερα αυτή η συγκυρία, ό,τι πολιτική και να κάνουμε, έχουμε ε, τον επιθυμητό πληθωρισμό, τον επιθυμητό σταθμισμό πληθωρισμό, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Οπότε, όπως είναι τα πράγματα, μας πανικοβάλλει αυτή η κατηφόρα που έχει πάρει η οικονομία. Άρα, τη γνώμη έχετε για τον όγκο του κυκλοφορούντος χρήματος, πώς είναι δυνατόν να έχει κάποια θετική επίδραση επί της απασχόλησης και κάτι άλλο. Πέστε μου δύο λόγια όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας της Ανατολικής Ευρώπης. Βέβαια, στα πλαίσια της σημερινής ε, δυσμενούς συγκυρίας. Βεβαίω, αυτό το οποίο ρωτάτε είναι πάρα πολύ εύστοχο και πάρα πολύ σημαντικό και όπως προείπα σε παγκόσμια κλίμακα, σε παγκόσμιο επίπεδο ζούμε μέρες αβεβαιότητας και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να προετοιμαστούμε. Το είπε η Κομισιόν. σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ιδέα ανάκαμψη θα γίνει όχι το 2009, το 2010. Δύσκολη χρονιά το 9. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Είναι σταθεροποίηση των προσδοκιών του πληθωρισμού, κάτι το οποίο είναι στοιχείο σταθερότητας ανάκτηση εμπιστοσύνη, άγγερα, θεμέλιο. Μείωση επιτοχίων, το οποίο βοηθάει τη μάχη του πληθωρισμού και οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη και σε δημιουργία θέσεων εργασία. Γι' αυτό το τελευταίο ζήτημα επαναλαμβάνω ότι η πρώτη δεκαετία του ευρώ όσον αφορά αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Χωρίς να υποτιμούμε τη δυσκολία της οικονομικής κρίσης, άρχισε πρόβλημα και με τα απασχόληση σήμερα. Δεν το λέμε αυτά ρίσκια, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτά, αυτό το, το μου της δεκαετίας. Εντυπωσιακό, μακρά περίοδος πετυχημένη νομίζω ότι πάνω από 3 εκατομμύρια 600.000 θέσει εργασία δημιουργήσαμε περισσότερες από ό,τι στις ε, είπα πολύ καλό για του Ευρωπαίους τώρα σχετικά αφορά τι δυνατότητε των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης νέων χωρών δεν νομίζω ότι μέσω μακροπρόθεσμα τους θίγει η κρίση, έχουν δυνατότητες. Φυσικά και η επιβράδυνση της ε, επηρεάζει, αλλά εάν συνεχίσουν οι χώρες αυτές τις ε, διορθωτικές μεταρρυθμίσεις τους που χρειάζονται, τότε οπωσδήποτε θα καλύψουν το χαμένο έδαφος και θα έχουν πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε τι γίνεται με τις τιμές βασικών εμπορευμάτων, καυσίμων, τώρα έχουν μειωθεί γιατί προηγουμένως ήταν πολύ ψηλές τιμές. Ήταν υπερβολικά ψηλές τιμές, τώρα ε, βρίσκονται στο άλλο άκρο και αυτό χωρίς να ε, Μπορείτε ποτέ να το υποτιμήσουμε. Ευχαριστούμε που τηρήσατε τα χρονικά μας ε, πλαίσια. Μένει ένα πεντάλεπτο. Catch the eye. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Προσέξτε, προσέξτε. Θα χρησιμοποιήσω εγώ το πεντάλεπτο. Ποιος θέλει το λόγο. Κοιτάξτε, εσεί δεν είσαστε μέλο της Επιτροπής. Ε, θα δώσω πρώτο λόγο στον κύριο Πέρβις. Ε, θεωρείτε ότι είναι πιθανό να υπάρξει κάποια αλλαγή λόγω και της αλλαγής της ε, κυβέρνησης στις ΗΠΑ, να υπάρξει κάποια αλλαγή σε επίπεδο κυβέρνηση, σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας. Κοιτάξτε, σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας η Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς, ε, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ε, και ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας παραμένουν τα ίδια άτομα. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Και πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε σημαντικές αποφάσεις Είχαμε κοινή απόφαση και με την ε, Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών ε, το γεγονός ότι ε, προσφέρουμε ρευστότητα σε δολάρια αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ στενή σχέση όπως σας είπα έχουμε τον εκτελεστικό βραχίωνα των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι σαφές ότι αυτή η αλλαγή της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά θεωρώ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ε, να ορίζουν το όραμά τους να έχουν τις δικές τους τις ε, αρχές. Πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε προετοιμασμένοι στο να είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να εξάγουμε τα μαθήματά μας από αυτά που παρατηρούμε. Και είναι αλήθεια ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε ε, να έχουμε με τη νέα κυβέρνηση μια εξίσου καλή σχέση ε, συμπεριλαμβανομένη και της επιτήρησης των πολιτικών. Κύριε Πρόεδρε, αν έπρεπε σήμερα να ισχύουν τα κριτήρια του Μάστριχτ, μήπως θα έπρεπε να προσθέσουμε και την σταθερότητα των χρηματο, χρηματαγορών. Είπατε, όλοι πιστεύουν βεβαίω ότι για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης ό,τι αφορά την εποπτεία θα αναλάβει αν θέλετε ξημένο ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επειδή πλέκονται και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργηθούν αν θέλετε απαραίτητε απαραίτητες γέφυρες. Τώρα όμως, υπάρχει αν θέλετε το «ή» αν θέλετε στο EMU που παρουσιάζει αν θέλει μια κάποια ισορροπία. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το M δηλαδή και σε ό,τι αφορά τώρα. Την, σε όλη την αντιμετώπιση τη κρίση, αγνοούμε δηλαδή την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση αν θέλετε των αποκαλωμένων φορολογικών παραδείσων. Με την Αμερικανική κυβέρνηση πιστεύετε ότι θα μπορέσει αν θέλετε να ενταθεί ο αγώνα αυτό και να βρούμε λύση στο πρόβλημα αυτό των φορολογικών παραδείσων. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σα παρατήρηση, θα έλεγα ότι όλε οι κεντρικέ τράπεζε παγκοσμίω αυτό θεωρούν ότι έχουν ε, μία ευθύνη. Έχουν ευθύνη σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Δεν σημαίνει βεβαίω αυτό ότι αυτή η ευθύνη θα πρέπει να τροποποιήσει την ίδια την νομισματική πολιτική. Διότι η επιχειρηματολογία που αναπτύσσουν οι κεντρικέ τράπεζε παγκοσμίω όλες οι θηγατρικοί φορείς, δηλαδή θηγατρικοί φορεί, λένε ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών είναι απαραίτητο στοιχείο, δηλαδή ικανή αλλά όχι αναγκαία. Γιατί δεν υπάρχει αντίθεση ε, στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και να αναλάβει επίση και την αναλότητα εξασφάλιση σταθερότητα των τιμών. Που όλε οι φορεί δηλαδή που στοχεύουν στην συγκράτηση του πληθωρισμού έχουν και έχουμε και εμεί στην Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή. Όλες οι κεντρικές ε, τράπεζες που γνωρίζω δημοσιεύουν τέτοιου είδου εκθέσεις σύνοπρα αφορά την σταθερότητα. Για να μπορέσουν να εκτιμήσουν και τους κινδύνους για τους οποίους θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν. Αυτό κάνουμε και εμείς βεβαίως στην Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή. Το περιβάλλον βεβαίως όλων των κεντρικών τραπεζών ως θεσμών είτε στην ομιλωτική ζώνη στην οποία ανήκουν, είτε στην χώρα του, είτε στην πολιτική ομοσπονδία, ή στη συνομοσπονδία τους, θεωρούνται ότι έχουν ε, αναλάβει ιδιαίτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την εξασφάλιση αυτής. Νομίζω λοιπόν πως το ερώτημα αυτό είναι θεμελιώδου κεφαλαιώδου σημασία. Δεν πιστεύω και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί η συνθήκη. Διότι να αλλάξει κανεί να τροποποιήσει μια συνθήκη ε, τη σήμερα ημέρα δεν είναι πράγμα εύκολο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αν θέλετε, παρουσιάζει το μεγάλο πλεονέκτημα το 105 έκτη παράγραφος. Ότι η τροποποίηση, αν θέλετε, έγινε εξ άντε. Και όλοι ξέρουν, ορισμένοι μπασπερτός, ξέρουν γιατί ομιλώ. Σε ό,τι αφορά το τώρα τελευταίο σα ερώτημα, το σχετικό με του φορολογικού παραδείσου αποκαλουμένους. νομίζω ότι ο όρο αυτό φορολογικού παραδείσου μου φαίνεται, αν θέλετε, πολύ. Έτσι, δεν λέει πολλά πράγματα. Μιλούμε για χρηματοοικονομικές αγορές δηλαδή που δεν σέβονται τους διεθνείς κανόνες σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη σταθερότητα των αγορών, τη διαφάνεια διαφάνεια των θεσμών δηλαδή αυτών των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αγορές δηλαδή που δεν ανταποκρίνονται και στους ε, κανόνες αν θέλετε στην ε, καταπολέμηση αν θέλετε του βρώμικου χρήματος, στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτοί ορίζονται διεθνώς και στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας. Εμείς είμαστε πολύ υπέρ της ενίσχυσης της εφαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο αυτών των κανόνων όπως ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι ίδιες οι έννοιες, δηλαδή εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Και το ίδιο ισχύει αυτό, αυτό σε αυτές τις αγορές δηλαδή. Η έννοια του φορολογικού παραδείσου είναι και κάπως σύνθετη. Γιατί Ακόμη και στην Ευρώπη οι φορολογίε δεν είναι ίδιε. Ακόμη και στην Ευρωζώνη η φορολογία δεν είναι ίδια, δεν είναι κοινή δηλαδή, εναρμονισμένη. Γι' αυτό λοιπόν όταν του αποκαλούμε φορολογικούς παραδείσους θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να ακολουθούν του κανόνε εποπτεία, ειλικρίνεια, ακαιρεότητα, α το πούμε έτσι, διαφάνειας, αν θέλετε, που αποτελούν αρχέ οι οποίες ισχύουν διεθνώς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ανταλλαγή, την τόσο μεστή και σημαντική ανταλλαγή απόψεων σε αυτή την χρονική στιγμή της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα έχουμε την ευκαιρία για να ξαναζητούμε για το τελευταία φάση του νομισματικού διαλόγου στις 30 Μαρτίου στο πλαίσιο αυτής εδώ της θητείας και ενδεχομένως τότε να κάνουμε και έναν απολογισμό της λειτουργίας αυτού του νομισματικού διαλόγου μέχρι τούδε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή και σας δίνω ραντεβού στις 30 Μαρτίου. Μη λυπεί ήδη η ιδέα ότι θα έχουμε το τελευταίο μας ραντεβού στις 30 Μαρτίου. Τέλη Μαρτίου, εν περιπτώσει, φέτος. Δεν ξέρω αν θέλετε τι κρίση, αν θέλετε θα επιφέρετε εσείς εδώ φορά τον νομισματικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς πάντως ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτές τις ε, δυνατότητες που μας δώσατε για να έχουμε αυτόν τον διάλογο μαζί σας. Και σας ευχαριστώ.